Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η Επιτροπή μας βέβαια δεν έχει συγκεντρωθεί ολόκληρη, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα σε όλους. Δεν είναι εδώ όλοι οι συνάδελφοι. Χθε όμως ήταν εντατική ημέρα. Κάποιοι λοιπόν μπορεί να βρίσκονται στα γραφεία τους. Να καλωσορίσω τον κύριο Γκαρίμπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια και τον κύριο Ζαμέ, Μέλο τη μέλος της ΕΣΡΕΚ. Είναι εδώ μαζί μα σήμερα για να σα παρουσιάσει μία μελέτη για την αμοιβαία αξιολόγηση προσωμιώσεων ακραίων καταστάσεων που διεξήχθησαν σε ευρωπαϊκούς πυρηνικού σταθμού. Δύο λόγια για να κάνω μια εισαγωγή σε αυτή τη σημαντική παρουσίαση, θυμίζοντα ότι η Επιτροπή μας μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα παρακολουθεί στενά το όλο θέμα της αξιολόγησης, της έκτασης μάλλον αυτού του γεγονότος και την ε, πραγματικότητα που επικρατεί στους πυρηνικούς σταθμούς της Ευρώπης. Ήδη τον περασμένο Ιούλιο είχαμε κάνει μια παρουσίαση από την ΕΝσρεκ για να αξιολογήσουμε μαζί με τους συμπερογνώμονες και τους εθνικούς φορείς την όλη κατάσταση στην Ιαπωνία. Το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας το λέω και στους προσκεκλημένους μας που το γνωρίζουν βέβαια, αλλά θέλω να το τονίσω, μας ε, αφορά άμεσα όπως με τις εκθέσεις μας έχουμε αποδείξει, με την έκθεση Μπρεζίνα λόγω χάρη για το πρόγραμμα Euratom ε, και το μέλλον του που επεξεργαζόμαστε με την έκθεση Skinner. Όλα αυτά στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή παρουσίαση δεν δείχνει απλώς το ενδιαφέρον μας για το όλο θέμα, αλλά είναι και συνέχεια μιας ε, διαδικασίας αξιολόγησης που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και στη διαδικασία λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή μας βάσει συγκεκριμένων εκθέσεων. Να δώσω λοιπόν το λόγο στους προσκεκλημένους μας, ευχαριστώντας τους για την προσέλευσή τους και την υπομονή τους, επειδή καθυστερήσαμε κάπως να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσετε εσείς, κύριε Γκαρίβα, με την πρώτη παρουσίαση. Σας ευχαριστώ, έχετε το λόγο. Δεν έχετε πολύ χρόνο, αλλά ξέρω ότι μπορείτε να είσαστε πολύ συνοπτικός. Σας ευχαριστώ. Uh, thank you very much, Mrs. President, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στις 25 Μαρτίου του 2011 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τρεις ε, υποχρεώσεις. Καταρχήν να αναπτύξει μια μεθοδολογία προκειμένου να διεξαχθεί ένας ε, εκτεταμένος, ε, μια εκτεταμένη αξιολόγηση μαζί με τις ε, ρυθμιστικές αρχές για τις προσωμιώσεις ακραίων καταστάσεων και μάλιστα να επεκταθούν αυτές οι δοκιμές σε όσο περισσότερες χώρες του κόσμου γίνεται στις γειτονικέ χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης να προταθεί αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια. Σήμερα θα ακούσουμε τον κύριο Ζαμέ από τη Γαλλική Αρχή Προστασίας και Ασφάλειας για το πώς έχουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την έκθεση εφαρμογής αυτών των προσωμιώσεων ακραίων καταστάσεων. Ο κύριος Ζαμέ ήταν πρόεδρος, εργαστικός πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου που επέβλεψε αυτή την αμοιβαία αξιολόγηση. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ όλους όσους άμεσα ή έμεσα έλαβαν μέρος στο έργο αυτό, γιατί πραγματικά ήταν μια δύσκολη και επίπονη χρονιά και σε λίγο χρόνο καταφέραμε σημαντικά αποτελέσματα. Οι μέχρι τώρα προσπάθειες ήταν αρκετά εντυπωσιακέ, ε, λαμβάνοντα υπόψη ότι το έργο αυτό έγινε σε οικειοθελή βάση από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα ήθελα να συνοψίσω τα τρία στάδια αυτή τη προσπάθεια. Καταρχήν, σε εθνικό επίπεδο. Ε, ύστερα από έτσι των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, οι φορεί όλων ε, και διαχειριστέ όλων των πυρηνικών σταθμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των άλλων δύο χωρών ε, τη Ελβετία και τη Ουκρανία που συμμετείχαν, ε, προέβησαν σε λεπτομερή έλεγχο των εγκαταστάσεών του με βάση τη μεθοδολογία που εκπονήθηκε και συμφωνήθηκε από όλε τι Ευρωπαϊκέ Ρυθμιστικέ Αρχέ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε εθνικό επίπεδο, οι ρυθμιστικέ αρχέ ανάλυσαν τι πληροφορίε και κατέληξαν σε εθνικέ ε, εκθέσει που δόθηκαν εμπρόθεσμα μέχρι την 31η δηλαδή Δεκεμβρίου του 2011. Οι αξιολογήσεις ξεπέρασαν ε, την τακτική αξιολόγηση προστασία που γίνεται στα πλαίσια τη ε, αδειοδότηση και των περιοδικών εκθέσεων. Αλλά θα ακούσουμε για αυτά τόσο λίγο. Βασικό στόχο είναι να ε, διδαχθούμε από τα παθήματα τη Φουκουσίμα και να εξετάσουμε το περιθώριο ασφάλειας ε, των Ευρωπαϊκών Πυρηνικών Σταθμών προκειμένου να καλυφθούν διάφορα περιστατικά και μάλιστα και συνδυασμό τους όπως συνέβη στη Φοκουσίμα με συνδυασμό του σεισμού και του τσουνάμι. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο περιεκτική αξιολόγηση των Ευρωπαϊκών Πυρηνικών Σταθμών και μάλιστα να γίνεται ταυτόχρονα με βάση τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές. Δεύτερο σημαντικό θέμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μία αμοιβαία αξιολόγηση έγινε μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του 2012 ενώ οι εθνικές εκθέσεις που προανέφερα από τις 17 συμμετέχουσες χώρες κάλυψαν πάνω από 150 πυρηνικού αντιδραστήρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αξιολογήθηκαν πάνω από 80 εμπειρογνώμονε από τι εθνικέ ρυθμιστικέ αρχέ 24 χωρών που είτε είναι πυρηνικέ δυνάμει είτε όχι. Και επίση συμμετείχε σε τη διαδικασία αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε και παρατηρητέ από μη κοινοτικέ χώρε, τον Καναδά, την Κροατία, την Ιαπωνία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τι Ηνωμένε Πολιτείε, καθώ και από την Διεθνή Υπηρεσία Ατομική Ενέργεια. Η αμοιβαία αξιολόγηση κατέληξε σε μια ενοποιημένη έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση με γενικές συστάσεις καθώς και 17 μεμονωμένες εθνικές εκθέσεις με λεπτομεριακές συστάσεις ανά χώρα και ανά πυρηνικό σταθμό. Όλες οι εκθέσεις αυτές βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΕΝΣΑ και μπορείτε να τις διαβάσετε αν το επιθυμείτε. Επίσης, στις 26 Απριλίου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, οι πυρηνικές ρυθμιστικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε κοινή δήλωση επισημένοντας την ανάγκη εκπόνησης ενός σχεδίου δράσης για να δοθεί μια συνέχεια στην αξιολόγηση που έγινε μέχρι τώρα και στο έργο που έγινε μέχρι τώρα και να εφαρμοστούν οι συστάσεις αυτής της αμοιβές αξιολόγησης από τις εθνικές αρχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει αυτό το σχέδιο δράσης μαζί με την ΕΝΣΡΕΚ στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει στις 3 Ιουλίου. Όταν θα συμφωνηθεί το σχέδιο δράσης και τα επιμέρους στοιχεία της εντολής του Συμβουλίου υλοποιηθούν, θα υποβληθεί ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, προκειμένου να λάβουμε και τις δικές σου απόψεις για, τη, για το τεστ αυτοαντοχής, τη διεθνή διάσταση, καθώς και το, τις γραμμέ γραμμές που θα ακολουθήσουμε μετά από την έκθεση αυτή και θα υποβάλουμε έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με βάση όλα αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που είσαστε και τόσο συνοπτικός, αλλά και τόσο σαφής. Και τώρα ο λόγος στον κύριο Φιλίπ Ζαμέ. Παρακαλώ. Merci beaucoup. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπατε, Είμαι ένα από του υπεύθυνου τη Εθνική Γαλλική Αρχή και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρισκόμαι μαζί σα σήμερα για να σας μιλήσω για τις ε, προσωμιώσει για τους πυρηνικού σταθμού της Ευρώπης και το πώς ε, παρακολουθήσαμε το θέμα. Είμαι υπεύθυνο λοιπόν για τα θέματα αυτά στην ε, Ευρώπη και, στη... και Γάλλος μεν πολίτης, αλλά θα είναι πιο δύσκολο για μένα να μιλήσω αγγλικά Ήθελα να κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Το τελευταίο που ήθελα να πω ότι προκειμένου να σας αφήσω και χρόνο για ερωτήσεις έχω αφαιρέσει κάποιες διαφάνειες από την παρουσίασή μου σε σχέση με αυτό που λάβατε ώστε να κερδίσουμε κάπως χρόνο και να υπάρξει περισσότερη συζήτηση. Θα περάσω στα αγγλικά. Η παρουσίαση μου λοιπόν διαιρείται σε τρία κεφάλαια. Ε, η σύνοψη τη διαδικασία των προσωμιώσεων και τη αμοιβέ αξιολόγηση. Μετά θα ανακεφαλαιώσω τα βασικά συμπεράσματα τη αμοιβέ αξιολόγηση και θα ολοκληρώσω με κάποια συμπεράσματα. Προτού περάσω στα ίδια τα τεστ της προσωμιώσης που έγιναν, να συνοψίσω τα βασικά διδάγματα του ατυχήματος της Φουκουσίμα, που ήταν βάση και για τη δική μας διαδικασία της αμοιβαίας αξιολόγησης. Τι μάθαμε δηλαδή και τι ερωτήματα αναγκάσαμε να θέσουμε στους εαυτούς μας με το ατύχημα αυτό. Πρώτον, όλα ξεκίνησαν με τον τεράστιο σεισμό και το τσουνάμι. Η φωτογραφία αυτή είναι φωτογραφία του πρώτου κύματος που πέρασε πάνω από την ε, από του Ταϊτσί. Μετά από αυτό βέβαια το κύμα όλο και μεγάλωνε και τελικά οι εγκαταστάσεις πλημμύρισαν τελείως. Εντός και εκτός με πολλές καταστροφές. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι ότι υπήρξε φυσική καταστροφή, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να προβλεφθεί σε τέτοια τοποθεσία. Δεύτερο στοιχείο το τεράστιο αυτό παλαιροϊκό κύμα και ο σεισμός μαζί κατέστρεψαν όλες τις ηλεκτρικές πηγές ενέργειας και το σύστημα ψήξης. Δηλαδή, όλα τα συστήματα ασφαλείας της, του εργοστασίου καταστράφηκαν ταυτόχρονα, ε, κατέστησαν ε, άχρηστα ταυτόχρονα. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι η κατάσταση εξελίχθηκε σε σοβαρότατο ατύχημα, πολλά ε, περιστατικά μαζί που δημιούργησαν ένα καταστροφικό ατύχημα, το οποίο δύσκολο μπορούσε κανεί να διαχειριστεί και βεβαίω δημιούργησαν και τα γνωστά προβλήματα διάξηση των περιβάλλων. Αυτέ είναι μερικέ από τι βασικέ πτυχέ του ατυχήματο, αλλά από την άποψη των προσωμιώσεων και τη αμοιβαία αξιολόγηση ε, θα, αναφέρω θα αναφέρομαι κυρίω αυτά τα τρία ζητήματα τα τρία ζητήματα που απασχόλησαν και τη διαδικασία τη αμοιβέ αξιολόγηση στην Ευρώπη για να δούμε και του εθνικού κινδύνου στην Ευρώπη, τα συστήματα ασφαλεία του και το πώ μπορούν να διαχειρίζονται τα εθνικά συστήματα, τα σοβαρά ατυχήματα. Πώ προχωρήσαμε τώρα, τι διαδικασία ακολουθήσαμε, η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε για την αμοιβαία αξιολόγηση και τι προσωμιώσει ε, ανα, αναπτύχθηκε από τη Βένρα. Η Βένρα είναι κάτι σαν ε, κλαμπ εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Εκείνοι είναι που από τεχνικής άποψης διευκρινίζουν πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτή η ομάδα υπέβαλε τις προτάσεις της, προτάσεις της στην ENSREG, ομάδα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή που, μας, που, εγκέκρι, που ενέκρινε τη διαδικασία για το πώς να προχωρήσουμε. Έτσι προέκυψαν λοιπόν οι τεχνικές προδιαγραφές. Ήδη ο Μάσιμο σας περιέγραψε τα διαφορετικά βήματα, δύο εθνικά στάδια και ένα τη αμοιβαία αξιολόγηση που συνδυάστηκαν. Θα ήθελα να επιμείνω στο εξή. Πολύ συχνά λέγεται ότι οι φορεί έκαναν μια αυτοαξιολόγηση και είπαν ότι ήθελαν. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Υπήρξε ε, μια έγκριση προδιαγραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά απαιτήθηκε από τους εθνικούς ε, ε, ζητήθηκε από του εθνικού φορεί με απέτηση των εθνικών ρυθμιστών να συμμορφωθούν με αυτέ τι απαιτήσει. Δηλαδή, οι εθνικοί ρυθμιστέ μπόρεσαν να ελέγξουν κατά πόσον έγιναν όσα απαιτήθηκαν και να ζητήσουν να επιβληθούν περισσότερα μέτρα ή να γίνουν περισσότερες βελτιώσεις. Μετά στην αμοιβαία αξιολόγηση εξετάστηκαν οι εκθέσεις που είχαν συνταχθεί από τους εθνικούς ρυθμιστές και το πώς αξιολόγησαν και τους φορείς και τις δικές τους τοποθετήσεις. Ανακεφαλαιώθηκαν λοιπόν όσο ήθελα να πω το πεδίο της αμοιβαίας αξιολόγησης ουσιαστικά εξέτασε τις εκθέσεις που είχαν συνταχθεί από τους εθνικούς ρυθμιστές και αυτό έγινε από εμπειρογνώμονες που όρισαν οι ρυθμιστές και από χώρε με πυρηνικούς σταθμούς αλλά και από χώρε χωρίς πυρηνικούς σταθμούς. Ήταν ανεξάρτητη λοιπόν αυτή η αμοιβαία αξιολόγηση από τους φορείς και από τους ρυθμιστές στην ουσία, αλλά δεν ήταν μόνο το κλαμπ των πυρηνικών χωρών, η ομάδα των χωρών με πυρηνικούς σταθμούς και οι ρυθμιστές τους που όριζαν αυτή τη διαδικασία. Οποιαδήποτε χώρα εκτός των χωρών με πυρηνικά εργοστάσια ήθελε να ορίσει εμπειρογνώμονα μπορούσε να το κάνει. Μάλιστα, οι εμπειρογνώμονες ήταν τελείως ισότιμοι. Είτε προέρχονταν από χώρες με πυρηνικούς σταθμούς είτε όχι. Κάτι άλλο που και ο Μάσιμο νομίζω ήδη το ανέφερε είναι ότι συμμετείχαν ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς πυρηνικούς σταθμούς, επίσης κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με πυρηνικούς σταθμούς, αλλά και παρατηρητές. Η διαδικασία τώρα της αμοιβαίας αξιολόγησης. Επί της ουσίας, η αμοιβαία αξιολόγηση διρέθηκε σε δύο βασικά στάδια στο πρώτο είχαμε να εξετάσουμε τις 17 εκθέσεις που είχαν συντάξει οι εθνικοί ρυθμιστές, όπως είχαν ετοιμαστεί δηλαδή στις διάφορες χώρες, και κατά πρώτον είχαμε μία έκθεση, μία ανακεφαλ... Ε, σύνοψη μάλλον ένα θέμα των εθνικών εκθέσεων, ζήτημα προς ζήτημα. Έπρεπε οι υπεύθυνοι να διαβάσουν τις εκθέσεις, να απευθύνουν ερωτήματα προς τους ρυθμιστές και να ετοιμάσουν είτε συνεντεύξει, είτε συνομιλίες και, συνεντε... συζητήσεις με τους εθνικούς ρυθμιστές. Αυτό ε, έγινε με 80 συμμετέχοντες. Κράτησε ένα μήνα η εξέταση των εκθέσεων στα γραφεία και επίσης υπήρξε και ένα εργαστήριο δύο εβδομάδων στο Λουξεμβούργο με 51, γύρ... με 51 γύρους συζητήσεων. Ήρθαν δηλαδή εμπειρογνώμονε, εξήγησαν τι έγινε για το καθένα από τα ζητήματα σε κάθε χώρα και απήντησαν σε ερωτήσεις που τέθηκαν από τους υπεύθυνου της αξιολόγηση. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος της αμοιβαίας αξιολόγηση. Δεύτερο στάδιο, η εξέταση κάθε χώρας από τους ε, ομότιμους εταίρους. Έξι ομάδες δημιουργήθηκαν, να επισκέφθηκαν τις 17 ε, χώρες που συμμετείχαν από 4-5 μέρες στην κάθε επίσκεψη. Σε αυτές τις επισκέψεις σε κάθε χώρα <clears throat> οι εμπειρογνώμονες και πάλι έθεσαν ερωτήματα από την πλευρά των ρυθμιστών ώστε να δουν περισσότερες λεπτομέρειες, να κάνουν προτάσεις ή κάποια πράγματα που είχαν παραβλέψει οι εθνικοί ρυθμιστές. Αυτό ήταν αρκετά δύσκολος διαδικασία. Επίσης οι επισκέψεις συμπληρώθηκαν από μία επίσκεψη σε εργοστάσιο που μπορούσε να επιλέξει κάθε ομάδα υπευθύνων. Κάποιες φορές προκαλείται σύγχυση στην όλη εικόνα για το πώς έγιναν οι επισκέψεις στα εργοστάσια. Δεν ήταν επιθεωρήσεις, δεν ήταν έλεγχοι. Δεν γίνεται επιθεώρηση έλεγχος από τέτοιες ομάδες. Απλώς έγιναν για να συλλεγούν ε, εντελεχείς πληροφορίες για το πώς ακριβώς είχε καταγραφεί η εικόνα κάθε στην έκθεση. Δηλαδή δεν ήταν αρκετό βάση των, του κάθε παραδείγματος να βρίσκονται όλα μόνο σε γραπτές εκθέσεις. Ένα σημαντικό στοιχείο της ε, έκθεσης ε, της ε, αμοιβαίας αξιολόγησης ήταν και η απήχηση στο κοινό. Να αναφέρω εδώ δύο βασικά στοιχεία. Υπήρξαν δύο δημόσιες ε, συναντήσεις ανοιχτέ για όποιον ήθελε να συμμετέχει. Πρώτη στις 17 Ιανουαρίου για την όλη διαδικασία της αμοιβές αξιολόγηση και επόμενη στις 8 Μαΐου μετά την ολοκλήρωσή της. Ώστε να δούμε τα πορίσματα. 200 περίπου ήταν οι συμμετέχοντε, μεταξύ των οποίων εθνικοί ρυθμιστές, με κυβερνητικέ οργανώσει, ε, το κοινό, φορεί και εκπροσωπή του και πολλέ φορέ υπήρξαν και φάσει ερωταπαντήσεων και συζήτηση. Έπειτα υπήρξε και ειδική σελίδα στον ιστότοπο τη ENSREG, όπου διατέθηκαν όλε οι εθνικέ εκθέσει και η αμοιβαία αξιολόγηση, με στοιχεία για τι προσημειώσει και τη διαδικασία τη αμοιβαία αξιολόγηση. Με τα οριστικά αποτελέσματα και πολλέ διαφάνειε, καθώ και διαρκή επικαιροποίηση του όλου εγχειρήματο. Έτσι μπορούσαν όσοι ενδιαφέρονταν να θέσουν ερωτήματα για την αμοιβαία αξιολόγηση. Τώρα, το αποτέλεσμα και η αποτίμηση της όλης διαδικασίας. Ε, μία βασική έκθεση που παρουσιάζει τα τελικά συμπεράσματα και τις συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα αυτό, ανακεφαλαιώνει την όλη διαδικασία, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μετά έχουμε και τις 17 αναχώρα εκθέσεις με πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα και συστάσεις που αφορούν την κάθε χώρα ξεχωριστά. Να συνοψίσω τα βασικά συμπεράσματα της ε, αμοιβαίας Δεν θα αναφερθώ στα συμπεράσματα αναχώρα βέβαια, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτο συμπέρασμα είναι ότι μετά την αμοιβαία αξιολόγηση είδαμε ότι έχουν αναλυθεί σημαντικά μέτρα σε όλες τις χώρες για να βελτιωθεί η ασφάλεια των εργοστασίων. Ο καθένα στην όλη διαδικασία τη αμοιβή αξιολόγηση και των προσωμιώσεων την πήρε πολύ σοβαρά. Αυτό φάνηκε από τα στα συμπεράσματά μα. Όμω, σίγουρο είναι ότι υπάρχουν κάποια θέματα με την επιμέρου ε, υλοποίηση ανάλογα με τα ρυθμιστικά συστήματα που διαφέρουν μεταξύ των χωρών στην Ευρώπη και βεβαίω ανάλογα και με την έκταση του κάθε πυρηνικού προγράμματο. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι υπάρχει γενικώ συνοχή στην Ευρώπη στο πώ εντοπίζονται τα καλύτερα χαρακτηριστικά τα ισχυρά σημεία του κάθε εργοστασίου, οι αδυναμίες και το τι πρέπει να βελτιωθεί ώστε να γίνει το κάθε εργοστάσιο πιο ασφαλές. Αυτό δεν ήταν δεδομένο από την αρχή. Μπορεί η ε, οπτική, σκοπιά και η μέθοδος αξιολόγησης να διαφέρει από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη. Δεν ήταν κάτι που το θεωρούσαμε σίγουρο. Όπως θα δούμε αργότερα όμως και στις συστάσεις, υπό ορισμένες σκοπιές υπάρχουν και αποκλήσεις. Γενικώ όμως λίγο πολύ υπάρχει και συνοχή. Και τελευταίο γενικό συμπέρασμα πριν τις συστάσεις μας είναι ότι σημαντικά μέτρα για να ενισχυθεί η ασφάλεια των εργοστασίων ή αποφασίστηκαν ή σχεδιάζονται στις περισσότερες χώρες. Πρόσθετος κινητός εξοπλισμός, λόγω χάρη ηλεκτρογεννήτριες ή αντλίες που θα μπορούσαν να προσθεθούν στο εργοστάσιο ή να μεταφερθούν εκεί εφόσον υπάρξει φυσική καταστροφή επιπλέον ακίνητο εξοπλισμό, σταθερό εξοπλισμό για την προστασία του συστήματος, εφόσον προκύψει κάποια φυσική καταστροφή, ας πούμε ένα σεισμός, αλλά και η διαχείριση των σοβαρών ατυχημάτων με την, ανάλογο, με την ανάλογη εκπαίδευση του προσωπικού. Αυτά διατίθενται ανά χώρα, σε κάθε μία από τις χώρες που βλήθηκαν σε έκθεση και σε εξέταση να καταλήξουμε τώρα στις τέσσερις βασικές συστάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που διατυπώνονται στην έκθεση. Η πρώτη αφορά την, τον καθορισμό των φυσικών ατυχημάτων, των κινδύνων και το τι μέτρα πρέπει να αναλυφθούν. Είπα ότι υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ έχουμε ένα από αυτά, μια από αυτές τις περιπτώσεις. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν την ίδια αντίληψη των φυσικών κινδύνων. Χρειάστηκε λοιπόν να γίνει και κάποια σχετική αποτίμηση και είδαμε ότι δεν υπήρχε συνέπεια από τη μια χώρα στην άλλη. Η πρώτη σύσταση της αμοιβαίας αξιολόγησης είναι ότι με την καλύτερη διαθέσιμη εμπειρογνωμοσύνη από όλη την Ευρώπη θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα σύνολο ορισμών για το τι εννοούμε με φυσικούς κινδύνους καθώς και την αξιολόγηση του περιθωρίου. Επίσης, η ανάγκη συστηματικής αξιολόγησης φάνηκε και πάλι από την όλη διαδικασία. Στις χώρες που συστηματικά υποβάλλονται σε πλήρη εξέταση των εργοστασίων, λόγω χάρη αναδεκαετία, στις χώρες αυτές, αναδεκαετία ακριβώς, Υπάρχει πλήρη εξέταση των εργοστασίων, των σταθμών και βλέπουμε αν αυτά τα εργοστάσια συμμορφώνονται με τι αρχικέ προδιαγραφέ ή κατά πόσον έχει βελτιωθεί η ασφάλεια. Ανάλογα με τι πιο πρόσφατε εξέλιξει, αυτό που φάνηκε από την αμοιβαία αξιολόγηση είναι ότι οι χώρε που συστηματικά υποβάλλονται σε έλεγχου είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και θέση να αποδείξουν ότι οι σταθμοί του είναι αρκετά ανθεκτικοί. Δεύτερη σύσταση λοιπόν, ΕΝΣΡΕΚ θα πρέπει να τονίσει τη σημασία ε, της συστηματικής αξιολόγησης ασφαλείας. Η τρίτη σύσταση έχει να κάνει με το ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας. Δείχνουμε εδώ κάποιες εικόνες από το τι είχε γίνει στη Φουκουσίμα αναλόγως. Να συνοψίσω το τι λέει αυτό το, αυτή η διαφάνεια. Το ατύχημα της Φουκουσίμα μας έδειξε τη σημασία να υπάρχει μια σταθερή δομή ε, αντιμετώπισης ώστε να μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τους ανθρώπους από τη ραδιενέργεια λόγω κάποιων ε, ατυχημάτων που έχουν προηγηθεί, όπως αυτό των 3 miles του 1979 Υπάρχουν κάποια στοιχεία που τα γνωρίζουμε ήδη πάρα πολύ καλά για το τι μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό που περάναμε από την αμοιβαία αξιολόγηση είναι ότι δεν μπορούν σε όλα τα εργοστάσια να υλοποιούνται όλα τα μέτρα με την ίδια ταχύτητα. Άρα, τρίτη σύσταση είναι ότι οι ρυθμιστέ θα πρέπει να σκεφτούν κατά πόσον μπορούν να απαιτούν την υλοποίηση όλων των μέτρων και αυτά να υλοποιούνται με ταχύτητα. Όσο το δυνατόν συντομότερα όποτε χρειάζεται. Τελευταία σύσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο Μάλλον, ένα από τα συμβιάσματα τη αμοιβέ αξιολόγηση ήταν ότι πρέπει να υλοποιούνται μέτρα για την πρόληψη των ατυχημάτων και την, τον περιορισμό των ε, επιπτώσεων του σε περίπτωση φυσικών κινδύνων. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούν και πάλι οι εθνικοί ρυθμιστέ. Για να είμαι λίγο πιο αναλυτικό, τι εννοούμε εδώ Πρώτον, αυτό είναι ένα άμεσο δίδαγμα του έλος από την περίπτωση της Φουκουσίμα. Οι ρυθμιστές θα πρέπει να απαιτούν από τους φορείς να είναι προετοιμασμένοι για καταστάσεις όπου υπάρχει πλήρης καταστροφή αλλά και απομόνωση του εργοστασίου, όπως στη Φουκουσίμα ακριβώς ή έπειτα περιστατικά με μεγάλη διάρκεια. Η κρίση στη Φουκουσίμα κράτησε αρκετέ εβδομάδε για να μην πω μήνε. Επίσης το να μην είναι διαθέσιμα αρκετά από τα συστήματα ασφαλείας, ξέρω, όπως η απουσία ηλεκτρικής ενέργειας ή οι αντλίες. Ακόμη να υπάρχει, αντλία, να υπάρχει μάλλον ε, απόθεμα ε, καυσίμων, Εφόσον πολλά ατυχήματα μπορούν να προκύψουν ταυτόχρονα σε κάποια εργοστάσια, αλλά να προβλέπονται και εκπομπέ ραδιενέργειε. Αυτό ήταν χαρακτηριστικό των όσων συνέβησαν στη Φουκουσίμα και έπρεπε να προπάρχουν μέτρα για να αντιμετωπιστεί τέτοια κατάσταση. Τέτοια μέτρα τα έχω αναφέρει όπως την, τον εξοπλισμό που έχει ήδη έχει ήδη προετοιμαστεί για αυτές τις περιπτώσεις κινητό εξοπλισμό, άμεση απόκριση, ομάδες διάσωσης με εξοπλισμό που είναι διαθέσιμος άμεσα. Λόγω χάρη κάποιοι που θα μπορούσαν να φτάσουν με ελικόπτερο στο εργοστάσιο. Ε, όσοι δουλεύουν ήδη στο εργοστάσιο μπορεί να είναι εξαντλημένοι. Υπήρξαν και κάποια θετικά στοιχεία που μάθαμε από την Φουκουσίμα. Το κτίριο που προστάτευε όσου εργάζονταν εκεί και μπορούσαν να, μείνουν μέσα και να προστατευθούν ακόμα και αν υπήρχαν εκπομπέ. Δεν ξέρω αν δεν υπήρχε αυτό το κτίριο κατά πόσο το εργοστάσιο θα είχε σωθεί σήμερα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαθέτουν όλοι οι σταθμοί στην Ευρώπη. Κάτι που θα πρέπει να σκεφτούν οι ρυθμιστέ για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πυρηνική κατάσταση. Για να ολοκληρώσουμε τώρα, η συνέχεια που θα δοθεί στην αμοιβή αξιολόγηση, νομίζω αυτή έδειξε ότι το να ανταλλάξουμε πορίσματα και συμπεράσματα από τις προσωμιώσεις μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών μπορεί μόνο να βελτιώσει την ασφάλεια και την αντεκτικότητα των εργοστασίων. Θα υπήρξουν και μελλοντικέ δράσεις που να προκύπτουν από τις προσωμιώσεις αυτές, οι οποίες σύντομα θα οργανωθούν από πρόγραμμα δράσης της ENSREG και οι οποίες θα συντονιστούν και με βάση τη σύμβαση για την πυρηνική ασφάλεια. Αυτά όλα τώρα σχεδιάζονται και στην, στις αρχές Ιουλίου θα υποβληθούν στην έντρη προς έγκριση. Ένα θέμα που θέλω επίσης να αναφέρω είναι ότι πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα και εκτός των εργοστασίων και επίγουσε καταστάσει, αλλά αυτό δεν βρισκόταν εντός της εντολής που είχε λάβει η Ένσφεγγ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Αυτό όμω είναι ένα από τα πρώτα μαθήματα που μάθαμε από τη Φουκουσίμα, γιατί υπήρχε μεγάλη ζήτηση που, να προκύπτει, που προέκυψε και από τις συζητήσει μα με το κοινό για το θέμα αυτό. Στο τελικό βασικό κεφάλαιο τη έκθεση, η αμοιβαία αξιολόγηση αναγνώρισε ότι η σημασία του να υπάρχει τέτοιου είδου ετοιμότητα στην Ευρώπη είναι σημαντικό. Είναι κάτι που θα πρέπει να το αντλήσουμε ω δίδαγμα από την καταστροφή τη Φουκουσίμα. Δύο ακόμη διαφάνειε και ολοκληρώνω. Καλά, πολύ γρήγορα. Η αμοιβαία αξιολόγηση ήταν μια πραγματική πρόκληση. Δεν θα το αναλύσω αυτό. Όταν ξεκινήσαμε δεν ήμασταν βέβαιοι ότι θα πετύχουμε. Απλώς πρέπει να πω ότι χρειάστηκε σημαντικός κόπος και δουλειά από 500 ε, τουλάχιστον εργαζομένους, από 150 μάλλον και να εξετάσουμε 150 αντιδραστήρες ανά την Ευρώπη. Ακόμη πρέπει να πω ότι η σκοπιά μας ήταν διεθνής εφόσον ασχοληθήκαμε το τι συνέβαινε στην Ιαπωνία και από εκεί παραδειγματιστήκαμε, αλλά και το τι συνέβαινε σε 17 χώρες της Ευρώπης, ανά χώρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. E- και εγώ θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που σας χειροκρότησαν, όμως επειδή πολλοί ζήτησαν το λόγο θα σας ζητήσω να είσαστε ε, σύντομοι, διότι στις 10 έχουμε σημαντικές ψηφοφορίες. Μάλιστα καθυστερήσαμε και λίγο, γιατί ήταν ε, πολύ λίγοι οι παρόντες, οπότε θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τώρα χρόνο. Η κυρία Σιζέλη. Ehm, ευχαριστώ, θα είμαι σύντομη πράγματι. Θα ευχαριστώ πολύ. Έγινε πολλή δουλειά. Η δε θέμενη αξία της ε, δουλειάς αυτής είναι στην ουσία μια προσπάθεια συγχρονισμού των εργασιών για την ασφάλεια. Απαιτούνται νέες αναλύσεις ξαναλέω ότι η προστιθέμενη αξία είναι ο συγχρονισμός των προσπαθειών για την εξασφάλιση της ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, στη βάση των αποτελεσμάτων, των συμπερασμάτων αυτών, αναμένεται να θεσπιστεί νέα νομοθεσία στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη δε βάση αυτή, να επέλθουν σημαντικές βελτιώσεις. Εγώ δεν τις έχω δει τις βελτιώσεις αυτές τις ουσιαστικές βελτιώσεις. Κάποιες βελτιώσεις υπάρχουν. Γι' αυτό ρωτώ, ποιες βελτιώσεις αναμένεται μετά από την ολοκλήρωση αυτών των stress test. Δεύτερη ερώτηση. Πρόκειται για θέμα εμπιστοσύνης βασικά. Μέχρι τώρα έχει, γίνει, έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό και το τεχνικό ε, τμήμα. Τι γίνεται με το πολιτικό τώρα κάποιος πρέπει να ενημερώσει, να διαφωτίσει την κοινή γνώμη για τα, το ποια ήταν τα συμπεράσματα των δοκιμασιών αυτών. Τελευταία, τρίτη ερώτηση μάλλον. Έχετε να πείτε κάτι για τις αρμοδιότητες των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και τις αντιδράσεις τους ευχαριστώ κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Ζαμέ για την παρουσίαση της αμοιβαίας αξιολόγησης. Είναι η δεύτερη φορά που παρακολουθώ τέτοιου είδους αξιολόγηση, αλλά και πάλι πιστεύω ότι είναι λίγο όριστη. Χαίρομαι που έγινε κάτι τέτοιο μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα, αλλά δεν έχουμε ένα φάσμα κριτηρίων. Και από τις 143, ε, από 143 πυρηνικούς αντιδραστήρες που έχουμε στην Ευρώπη, ποιοι είναι οι πιο επικίνδυνοι, ποιοι είναι τα πιο επικίνδυνα πυρηνικά εργοστάσια που χρειάζονται κατεπηγόντως κάποιες εργασίες επιδιόρθωσης, ενώ ποια, ποια άλλη πυρηνική σταθμή ανταποκρίνονται σε ε, υψηλέ προδιαγραφέ ασφάλεια. Μια οριστή επικρατή. Μιλήσατε για επιθεώρηση αναχώρα. Αλλά ε, σε άλλε χώρε έχουμε τρει μόνο πυρηνικούς σταθμούς. Ε, στην Γαλλία έχουμε 100 και... 58. Συγγνώμη, στην Γαλλία έχουμε 58 σταθμούς πυρηνικούς. Πώς γίνεται αυτή η επιθεώρηση. Επίσης μιλήσατε για τον πυρηνικό σταθμό του Φεσολνάιν. Είπατε ότι ίσως ε, δημιουργηθεί μόλυνση στον υδροφόρο ορίζοντα. Επίσης είπατε ότι ε, αίθουσε ελέγχου που είναι ανεξάρτητε από τι αίθουσε ελέγχου εντό του πυρηνικού σταθμού. Τι χρονοδιάγραμμα έχετε προβλέψει για τα έργα αυτά που απαιτούνται και τι αξιολόγηση του κόστου γίνεται. Γιατί είπαμε τι θα γίνει με τον ορίζοντα Ευρώπη 2020 για την πράσινη οικονομία. Υπάρχει ένα υπολογισμό του κόστου για όλε τι εργασίε αυτέ που είναι απαραίτητε. Και τι γίνεται με την υπεργολαβία. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαμε στη Φουκουσίμα αλλά και σε άλλε χώρε είναι το πρόβλημα των υπεργολάβων που μπορεί να είναι 7 διαφορετικά επίπεδα και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε επίπεδο ασφάλειας και προστασίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαντό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι οι οικολόγοι θέλουν εξάλληψη του πυρηνικού κινδύνου και δίνουμε μάχη για να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο κίνδυνος από τα πυρηνικά. Εγώ θα ήθελα να μας υπενθυμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τα τεστ αυτά αντοχής ουσιαστικά σηματοδοτούν μια αποτυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια ήττα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο της 25ης Μαρτίου οι Υπουργοί ζήτησαν εξονυχιστική και ευρυθή ανάλυση του κινδύνου από τα πυρηνικά εργοστάσια και μόνο με την πίεση της ΕΝΣΡΕΚ και της ΟΥΝΡΑ έγιναν αυτά τα τεστ και μάλιστα επικεντρώθηκε σε θέματα σεισμικών κινδύνων και πλημμυρών. Και θυμάμαι ότι ο Επίτροπος Έτιγκερ ε, ουσιαστικά αναγνώρισε την πολιτική του ΙΤ απέναντι στην ΣΡΕΚ και την ΟΕΡΑ. Έχουμε μια καλή άσκηση μεθοδολογίας και επικοινωνίας όπως μας είπατε, αλλά θα έλεγα, συνοψίζοντας, Κάτι που έλεγε ο ο πρώην, επίτροπος, ο πρώην πρόεδρος της ε, Γαλλικής Δημοκρατίας, ο κ. Σαρκοζή, Σαρκοζή ότι δεν θα έχουμε στο Φενσενάιμ Φουκουσίμα γιατί δεν πρόκειται να φτάσει Παλιριακό και είμαστε στην περιοχή αυτή. Έχουμε όμως ε, διάφορους ε, κινδύνους από ανθρώπινα, τεχνικά λάθη, δολιοφθορά και το συνδυασμό των διαφόρων παραγόντων που επίσης προκαλούν σημαντικά πυρηνικά ατυχήματα και δυστυχώς ε, δεν αναλύθηκαν αυτά στα, στις προσωμιώσεις ακραίων καταστάσεων. Μετά τη Φουκουσίμα περιμέναμε ότι ο κίνδυνος ε, σημαντικών ατυχημάτων θα εξεταζόταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φαίνεται ότι περιοριστήκαμε μόνο στην ανάλυση του σεισμικού κινδύνου ή του κινδύνου πολυεργικού ε, κύματος που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους Ευρωπαϊκού πυρηνικού σταθμού. Αυτό είναι απαράδεκτο για μας και ανεπαρκές, γιατί θα πρέπει να καλύψουμε ένα πολύ ευρύτερο ε, φάσμα κινδύνων. Ο κύριο ε, Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι Λιθουανός και βέβαια με ενδιαφέρει το θέμα και πολλές από τις πτυχές του αθέματος που ακούσαμε σήμερα. Πολλές συζητήσεις γίνονται τώρα για τους μελλοντικού πυρηνικούς σταθμούς που πρόκειται να οικοδομηθούν, να κατασκευαστούν. Και βέβαια ανακύπτουν και πολλά ερωτήματα σχετικά με τους αντιδραστήρες των εργοστασιών αυτών. Γνωρίζετε ότι η Λιθουανία ακόμη δεν έχει παροπλήσει τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της. Διερωτώ με εάν η Κομισιόν διαθέτει σχέδια σχετικά με την αξιολόγηση των ε, αντιδραστήρων που βρίσκονται σε χρήση σήμερα και αν μετά από τις δοκιμασίες αντοχής έχει καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με το ποιοι από τους αντιδραστήρες αυτούς θα πρέπει να κλείσουν γιατί δεν είναι ασφαλής. Επίσης αυτές οι επισκέψεις των 4 ή 5 ημερών βρίσκω ότι είναι πολύ σύντομες και αμφιβάλλω αν αξίζουν τον κόπο γιατί τα πράγματα που μαθαίνουν οι εμπειρογνώμες μπορούν να τα μάθουν και από τη γραπτή τεκμηρίωση. Είπατε ακόμη ότι μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας εξαρτώνται από τις διαθέσεις των ηγεσιών των χωρών μελών. Μπορείτε να μας πείτε ποιες είναι οι χώρες εκείνες μέλη οι οποίες δεν έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα της πυρηνικής ασφάλειας. Και τέλος, για το θέμα της προστασίας των προστατευτικών περιβλημάτων. Αυτό σημαίνει βέβαια τεράστια επένδυση. Εφόσον δηλαδή δαπανώνται τόσα κονδύλια, τόσα χρήματα για να κατασκευαστούν τα προστατευτικά αυτά περιβλήματα και να ενισχυθούν κτλ. Αυτό σημαίνει ότι τελικά είναι υπερβολικά δαπανηρή η ε, πυρηνική ενέργεια. Η Ρεβέκα, κυρία Χάρμς, πρώτα θέλω να θέσω το ερώτημα. Εάν τα stress test έχουν ολοκληρωθεί, διότι την τελευταία φορά που ήρθε εδώ ο Επίτροπος Oettinger και τον ρωτήσαμε για το θέμα αυτό, μας δήλωσε ότι θα είναι απαραίτητες και άλλες επισκέψεις σε τέσσερα πυρηνικά εργοστάσια. Τρία από αυτά είπε ότι ήταν το Φέσενχάιμ, Τέμεριν και Κατενού. Δεν είπε ότι ήταν το τέταρτο εργοστάσιο. Θα ήθελα να μάθω εάν οι επισκέψεις αυτές όντως θα διεξαχθούν ή εάν εκεί ο Επίτροπος μας είχε ανακοινώσει κάτι το οποίο εν τέλει δεν έχει τεθεί ως θέμα στην συζήτηση αυτή περί stress test και επίσης ποιες είναι οι αναγκαιότητες επανεξέτασης στις επισκέψεις αυτές. Και συμπληρώνοντας αυτό που ερώτησε ήδη η συνάδελφός μου, ερώτησε σχετικά με αυτό το second containment, το δεύτερο προστατευτικό περίβλημα. Γιατί δεν έχει εξεταστεί, και ρητά μάλιστα μας το λέτε αυτό, γιατί δεν διερευνήθηκε ποια, εργοστάσια είναι καλύτερα, ποια είναι λιγότερο καλά. Μιλήσατε για το προστατευτικό περίβλημα μόλις στο τέλος της ομιλίας σας. Τώρα θέλω περισσότερες διευκρινήσεις και ιδίως εάν πρόκειται να γίνουν και άλλες έρευνε έρευνες σε σχέση με τον ενδεχόμενο κίνδυνο πτώσης αεροσκάφους. Εγώ επισκέφθηκα την Ιαπωνία προ λίγων μηνών και γνωρίζω ότι ο έλεγχος δεν εξασφαλίστηκε μετά από λίγες εβδομάδες. Ακόμη σήμερα δεν είναι, δεν είναι υποέλεγχο οι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Ακόμη μέχρι σήμερα προσπαθούν να αναπαραστήσουν, να ε, καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με το πώς έγινε το ατύχημα, πώς εξελίχθηκε το ατύχημα. Και αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η διαχείριση της καταστροφής. Τρεις αντιδραστήρες ταυτόχρονα και το σενάριο αυτό της διαρκούς απελευθέρωσης στο φυσικό περιβάλλον τεράστιων ποσοτήτων ραδιενέργειας μέχρι τώρα το σενάριο αυτό δεν έχει τεθεί ως βάση των ε, μελετών μας. Η εκένωση του Τόκιο που συζητήθηκε τι σημαίνει αυτό ως ενδεχόμενο για τα μεγάλα αστικά κέντρα που βρίσκονται στην Ευρώπη κοντά σε ε, πυρηνικά ε, εργοστάσια. Για παράδειγμα το Παρίσι ή για παράδειγμα οι Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ακόμη τέσσερις ε, παρεμβάσεις και θα έχουμε 7 λεπτά για την απάντηση. Ένα λεπτό καθένας παρακαλώ, γιατί έχουμε και ένα τέταρτο καθυστέρηση στην αρχή. Σας παρακαλώ να είστε συνεργάσιμοι. Και ευχαριστώ και για την παρουσίαση. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, δεν θεωρείτε ότι η βασική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η πλήρης εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας και μάλιστα από όλα τα κράτη-μέλη. Πόσα κράτη-μέλη μέχρι στιγμής έχουν ενσωματώσει στην ένωμη, στην του τάξη την οδηγία ε, για την ασφάλεια που κανονικά από τον Ιούλιο του 2011 έπρεπε να έχει εφαρμοστεί. Και αυτά τα τεστ αντοχής μήπως ε, είναι εξαίρεση στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή πύρο. και τι ρόλο θα παίξουμε στην εναρμόνιση των προδιαγραφών ασφάλειας αλλά σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φράγκο. Κυρία Χολ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζαμέ για την ε, τόσο σαφή παρουσίαση. Απλώς ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο που το θίξατε κι εσείς. Το θέμα της απομόνωσης. Τι γίνεται εάν ένας πυρηνικός σταθμός αποκοπεί είτε γιατί το εργοστάσιο αυτό ξαφνικά έχει μολυνθεί, είτε γιατί η επικοινωνία, η διασύνδεση με το εργοστάσιο ε, από ξηράς δηλαδή οδοί και τηλεπικοινωνίες επίσης έχουν διακοπεί. Με ανησυχεί, ανησυχεί κάπως ότι δίνεται έμφαση στον κινητό εξοπλισμό, το προσωπικό που θα πρέπει να μεταφέρεται έξωθεν. Αυτό δεν θα μπορεί να λειτουργήσει ένα απομονωμένο και αποκομμένο ένα εργοστάσιο. Πιστεύετε λοιπόν ότι γίνονται αρκετά στα παθητικά συστήματα ασφαλεία. Πώ γίνεται να είναι αντιδραστήρε ασφαλή, εάν ξαφνικά δεν μπορεί να έρθει και βοήθεια από έξω. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι χώρες που ήδη διαθέτουν πυρηνικού σταθμούς βρισκόνται σε διαφορετική θέση από αυτές που τώρα χτίζουν τα εργοστάσια τους. Η Πολωνία, λόγω χάρη, αυτή τη στιγμή κατασκευάζει πυρηνικό σταθμό. Τα νέα πρότυπα ασφαλείας βεβαίως και θα επηρεάσουν το κόστος κατασκευής. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω πότε θα αποστείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λεπτομερείς πληροφορίες για τις απαιτήσει ασφαλείας με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι νέοι πυρηνικοί σταθμοί. Σας ευχαριστούμε κύριο Σκίνερ. Σας ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που δεν παρακολουθήσα ολόκληρη τις παρουσιάσεις. Όμως ήθελα να ρωτήσω το προσωπώση. Δηλαδή Η γεωγραφική τοποθεσία ήταν κριτήριο κατά την εξέταση στις προσωμιώσεις. Δηλαδή η πιθανότητα σεισμού ή παλιολογικού κύματος στην Ευρώπη σε πολλές γεωγραφικές τοποθεσίες δεν είναι τόσο μεγάλη πιθανότητα. Άρα ανακουφίστηκαν και διασκεδάστηκαν ησυχίες ή το αντίθετο. Βεβαίω, ε, η διαδικασία αξιολόγηση είναι σε εξέλιξη και καλό είναι να υπάρχει και ευαισθητοποίηση για το θέμα τη πυρηνική ασφάλεια. Αλλά εάν θέλουμε να βασιζόμαστε σε χειροπιαστά δεδομένα, ε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν. για τα ε, αεροσκάφη. Κατά πόσον θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τέτοιες ε, καταστάσεις. Bene, abbiamo moltissime domande e 3-4 minuti. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και 3-4 λεπτά για την απάντηση από τον κύριο Γκαρίμπα και τον κύριο Ζαμέ. Θα προσπαθήσετε εσείς να περιοριστείτε. Ευχαριστώ. πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που τέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κύριος Ζαμέας απαντήσει στα πιο τεχνικά θέματα που ε, ρώτησαν οι ευρωβουλευτές. Πρώτα, σημείωσα ότι ορισμένες ερωτήσεις αναφέρονταν σχετικά σε, μάλλον αναφέρονταν σε νέα νομοθεσία για την πυρηνική ασφάλεια. Κοιτάξτε, Πώ κινούνται διαδοχικά τα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συντάξει έκθεση που θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίω, η οποία έκθεση προβλέπεται για τον επόμενο Οκτώβριο. Μετά ελπίζουμε ότι θα διεξαχθεί πλήρη συζήτηση που θα προχωρήσει μετά στην υποβολή της σχετικών νομοθετικών προτάσεων. Οι περιοχές που θα κινηθεί νομοθεσία θα είναι η διαχείριση, governance δηλαδή, από πλευρά των ε, εθνικών αρχών. Δεύτερον, τεχνικά κριτήρια που θα ενσωματωθούν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και τρίτο, πώς να βελτιωθεί η διαφάνεια στον ε, πυρηνικό τομέα. Ορισμένες ερωτήσεις τέθηκαν γύρω από τα θέματα ασφαλείας. Η ομάδα εργασία του Συμβουλίου για την Πυρηνική Ασφάλεια έχει δώσει τελική μορφή στο έργο της και το δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου. Άρα, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εξετάσετε το κείμενο εκεί. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τις απόψεις της όταν θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μία ερώτηση τέθηκε ακόμη σχετικά με το καθεστώς των stress test. Βρίσκω ότι είναι σημαντική ερώτηση αυτή με την έννοια ότι κάτι που είναι απολύτως θεμελιώδες είναι τα αποτελέσματα των δοκιμασιών αντοχής να εφαρμοστούν ορθά από τις εθνικές αρχές. Πάνω σε αυτό εργάζονται εθνικοί ρυθμιστές και Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα δημοσιεύσουμε το σχέδιο δράσης μας. Ελπίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα και τα τεχνικά θα απαντήσει ο Φιλίπ. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι πιο τεχνικό αυτό που θα πω τώρα. Υπενθυμίζω κάτι το οποίο απασχόλησε πολλούς παρεμβάντες. Η ευθύνη για τον έλεγχο και την ασφάλεια παραμένει εθνική αρμοδιότητα των εθνικών ρυθμιστών. Και αυτό έχει σχέση και με τις επιτόπου επισκέψεις. Δεν με ακούτε? Σας ακούω, λέει η κυρία Χάμς. Εγώ αναμένω απάντηση από την Κομισιόν για το πρόγραμμα των επισκέψεων. Δυστυχώς μιλούν. Επαναλαμβάνω, την ευθύνη φέρουν οι εθνικοί ρυθμιστές. Εγώ θα τρόμαζα εάν όλη την ευθύνη την αναλάμβαναν οι επισκέψεις αυτές των 4-5 ημερών. Η ευθύνη λοιπόν δεν μπορεί να γίνει με τον τρόπο αυτό, να αναλυθεί με τον τρόπο αυτό. Δεν είναι επιθεωρήσεις, είναι επισκέψεις ενδιαφέροντος, α το πω έτσι. Τώρα, το κόστος των μέτρων, μπορώ να απαντήσω για τη Γαλλία, το, το κόστος για κάθε σταθμό είναι μεταξύ 100 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα άλλο τεχνικό θέμα είναι, δεν μπορεί να πει κανείς ότι το στρες έγινε μονάχα για φυσικές καταστροφές. Βεβαίως το πρώτο θέμα ήταν αυτό, θεομηνίες και φυσικές καταστροφές. Αλλά λάβαμε υπόψη και άλλους παράγοντες και το management πώς θα γίνει και για άλλους κινδύνους. Έχουν ολοκληρωθεί τώρα τα stress test, όπως είπε ο Μάσιμο. Βρισκόμαστε στην φάση εφαρμογής και ε, του να καταστούν γνωστά τα αποτελέσματα. Η πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τις απαντήσεις σας και κάποιες πιο λεπτομερείς θα τις ακούσουμε φαντάζομαι σε άλλες ευκαιρίες που θα έχουμε να συναντηθούμε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την παρουσίαση της μελέτης και ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν. Ας περιμένουμε λίγα λεπτά για να καθίσουν όλοι και μετά προχωρούμε στις ψηφοφορίες.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 Εάν είναι έτοιμοι οι συνάδελφοι να ξεκινήσουμε και παρακαλώ όσοι δεν θα συμμετάσχουν στις προφορίες ας φύγουν. Να ξεκινήσουμε. Έφτασαν οι κατάλληλοι. tutti eh? όλοι, κύριε Βιντάλ Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα να δούμε αν λειτουργούν τα μηχανήματα. Και αν είναι σωστά, σωστή αριθμή των βουλευτών. Όποιος θέλετε λοιπόν να γίνει σωστά ο έλεγχος, ψηφίστε ναι. Είμαστε όλοι εδώ, ψηφίσατε. Ancora qualcuno Κάποιοι δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Οκ. Votazione chiusa. Πέρας της ψηφοφορίας. Κάποιος ψήφισε κατά του εαυτού του. Κάποιος ψήφισε όχι. Λοιπόν, θα σας ζητήσω εδώ τη συνεργασία σας γιατί να με ο κατάλογος των ψηφοφοριών και σε κάποιε περιπτώσει είναι και κάπως περίπλοκες οι ψηφοφορίες. Λοιπόν, ας είμαστε όλοι συνεργάσιμοι, να σηκώνετε οπωσδήποτε τα χέρια. Πρώτη έκθεση του κυρίου Κάριον που συζητήσαμε χθε. Θα ψηφίσουμε για το κείμενο ε, μετά τις διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, το συμβαστικό κείμενο, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Votazione aperta. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντε. Ένα βουλευτή του ΕΛΚ είναι υπεράριθμο. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι. Και πάλι έχουμε ένα παραπάνω από το ΕΛΚ. Σας παρακαλώ, βγάλτε την κάρτα από το μηχάνημα αυτός που πλεονάζει. Εψήφισαν άπαντες, εγκρίνεται. 36 προς 18 εγκρίθηκε. Πρέπει να ψηφίσουμε για το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato άπαντες, πέρας. Και πάλι ένας βουλευτής του ΕΛΚ παραπάνω. Avete votato tutti, votazione chiusa, è approvato. εγκρίθηκε το ψήφισμα. Votazione chiusa. Complimenti al collega Karinz. E Συγχαρητήρια στον κύριο Κάριντς. Δεύτερη ψηφοφορία. Πρόταση κανονισμού για την περιφερειακή ανάπτυξη. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Εντάξει. 52. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Εγώ θα το κάνω. Παρακολουθήστε με. 52. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 52. Ε, 52, ναι. 52. Εψήφισε να παντές πέρας. Πέρας. Απορρίπτεται. Πενήντα τρία. Όχι, με συγχωρείτε. Τρία. Τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πενήντα τρία. Καταπίπτει. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πενήντα επτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Έξι υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμμεβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε για να είναι σίγουρο. 62. Ένα σοσιαλιστής τώρα πλέον να ζει. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν ψήφισαν άπαντες. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Νομίζω ίδια πλειοψηφία με πριν. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικός. Για την 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 να το ελέγξουμε και αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Ψήφισαν όλοι. Κάποιος λείπει. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. 66. 66. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο. 66. Ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 68. Υπέρ. Καταβίπτει, καταβίπτει 67. Πιλάρ. Όταν, 60, εφόσον 66 εγκρίθηκε, 67 καταβίπτει. 68 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Λείπουν κάποιοι. Πέρας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 69 καταπίπτει. 70. 70. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 71 και 72. Πανομοιότυπος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβεβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81 Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 15 καταπίπτει. 82. Καταπίπτει και αυτή. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά σε ελέγξουμε. Κοιτάξτε, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε μία και δύο ψήφους διαφορά, οπότε καλύτερα να ελέγξουμε. 84 λοιπόν, ε, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται.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 κατά, αποχές εγκρίνεται, 91 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 92 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 93 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Έλεγχο, όχι έλεγχο. Για το 97 έλεγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πάλι ένας ε, του ΕΛΚ υπεράριθμο. Παρακαλώ βγάλτε την κάρτα σα. Πέρα. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά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 Εγκρίνεται. 35, 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε για, τον, για την 106. 106. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται.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 αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 37 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ, κατά, αποχές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 Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. Σαράντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σαράντα ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Άρχεται την ψηφοφορία για την τροπολογία 41. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται με δύο ψήφου διαφορά. Με συγχωρείτε, αλλά κάποιε φορέ είναι δύσκολο. Με μία-δύο ψήφου διαφορά, πού να καταλάβει κανεί. Και δεν είναι και όλε οι ομάδε πλήρε. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται, συγγνώμη. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται η ψηφοφορία Avete votato tutti? La votazione è chiusa. Peras. Εγκρίνεται η έκθεση. Με μεγάλη πλειοψηφία. Περνάμε τώρα, μετά το πέρας της προφορίας φυσικά, στον γενικό κανονισμό με την κοινή θέση για τα ταμεία. Είστε έτοιμοι? Εδώ Έχουμε κατάλογο ψηφοφοριών, το γνωρίζουν οι σκιώδεις εξηγητές, κατάλογο ψηφοφοριών με ομάδες τροπολογιών όταν είναι παρόμοιο το περιεχόμενο. Όταν λοιπόν ψηφίσουμε μια τροπολογία, ισχύει αυτό για το σύνολο των τροπολογιών. Ξεκινούμε με την τροπολογία 49. Καλύπτει όλα τα άρθρα στα οποία υπάρχει παραπομπή άρα και τις ε, σχετικέ ψηφοφορίες. Θα ήθελε να ψηφίσουμε όμως ηλεκτρονικώ για την τροπολογία 49, άρχεται η ψηφοφορία. 49, η Τροπολογία 49, άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν άπαντε. Λείπει Κάποιο, πέρα. Απορρίφθηκε. Η 49 απορρίφθηκε, άρα και όλες που βρίσκονταν στην ίδια ομάδα για τις περιοχές μετάβασης. 50. Και εδώ έχουμε ψηφοφορία σε ομάδα. Δηλαδή 81, 89 και ούτω καθεξής που αφορούν τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και εδώ να ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς για να είμαστε βέβαιοι. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 50, ε. Για, το, για την ομάδα της 50. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίθηκε. Άρα εγκρίνεται και η 50 και οι υπόλοιπε της ομάδας της. Δεν θα τις ψηφίσουμε. Εγκρίθηκαν τώρα. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Παρακαλώ, για να συντομεύουμε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 53 απορρίπτεται. 54 πάλι ομάδα με τις υπόλοιπες τροπολογίες υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 54 και οι υπόλοιπε δικές της. 55. Θέλετε έλεγχο για την 54, παρακαλώ. 54 με την ομάδα της ε, έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Χαρήκατε κυρία Τσίτσεστερ. 55 και λοιπές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. 55. Votazione aperta, Εψήφισαν άπαντες. Υπάρχει πάλι ένας πλενάζων από το ΕΛΚ. Παρακαλώ βγάλτε την κάρτα σας. Εψήφισαν άπαντες. Πέρασε. Εγκρίνεται. Οι 55 και εγκρίθηκαν. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 και λοιπές. Μεγάλη ομάδα τροπολογιών. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 59 και λοιπές. Η 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65 καταπληκτή. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Εγκρίθηκε. Καλά έλεγχος. 67. Ας επαληθεύσουμε. Ηλεκτρονικός, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 69. Άρχεται η ψηφοφορία. να άπαντες. Πάλι ένα από το ΕΛΚ παραπάνω. Βγάλτε το μηχάνημα παρακαλώ. Το, την κάρτα από το μηχάνημα. Πέρας. Απορρίπτεται με δύο ψηφού διαφορά. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 86 συγγνώμη 86 υπέρ κατά αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 86, άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι πλεονάζει ένας. Βγάλετε παρακαλώ την κάρτα σας, πέρας. Εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 91 chi è 91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Για να αποφύγουμε ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. 93 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν ανάπαντες. Πάλι ένας του ΕΛΚ είναι υπεράριθμος. Πέρας. Εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 97 συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 πάλι σε ομάδα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 και λοιπές. 104 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 100 καταρρύπτουν όλες. Όλες οι επόμενες καταρρύπτουν και φτάνουμε στην 111 ε, ομάδα με τις υπόλοιπες Υπέρ. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 119. 119, ναι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. 122. 122. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λάμπερτ. Άρχεται η ψηφοφορία. Είτε votato tutti. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Με μία ψήφο διαφορά απορρίπτεται. 123. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 124. Ηλεκτρονική ψηφοφορία Λάμπερτ. Για να είμαστε βέβαιοι. 124. Εψήφισαν άπαντε. Πάλι λείπει κάποιο. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Απορρίπτεται. 125. Λάμπερτ ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ε, απορρίπτεται συγγνώμη. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Έλεγχος. Κάποιοι θέλουν να ελέγξουμε. 155 ψηφίζουμε ηλεκτρονικός. Vi prego di votare. La votazione è chiusa. Εγκρίνεται. 156. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικός απευθείας για να είμαστε βέβαιοι. 156. Άρχεται η ψηφοφορία. 156. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 158. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 159. ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ εποχές εγκρίνεται. Έλεγχος, έλεγχος για την 166. 166, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία. 28 προς 28 απορρίπτεται. 167. 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θεωρώ ότι απορρίφθηκε. Έλεγχο. Ας κάνουμε έλεγχο για την 181. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Κάποιος λείπει. Πέρασε. Εγκρίνεται με δύο ψηφούς τη φορά. Ε, 183 ή 182 καταπίπτει. 183. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν αρχεται ψηφοφορια εψηφισαν Πέρας. περά. εγκρινεται 184 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 187 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ας ελέγξουμε 187 έλεγχος Εψήφισαν άπαντες. Πέρας της ψηφοφορίας. Μία ψήφος διαφορά. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 191. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 196 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 197 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 198 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 201. 201 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε για την 201. 201, ηλεκτρονική ψηφοφορία. E άρχεται η ψηφοφορία και πέρας. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. 202. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 200 έλεγχος. Για την 202 ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία. Avete votato tutti? Il voto è Εψήφισαν άπαντες, πέρας. Εγκρίνεται. 204. Ηλεκτρονική ψηφοφορία απευθεία. Για να είμαστε βέβαιοι. 204. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. 205. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν Πέρας. Εγκρίνεται. 209. 209 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 210 ηλεκτρονική ψηφοφορία. 210 ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 211 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 212 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 ηλεκτρονική ψηφοφορία. 214 εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά αποχές 216 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 219. 219 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 219. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 220 καταπίπτει. 221. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 222. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 225. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 226 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 220, 230 μάλλον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 233 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 234 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 235 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μου φαίνεται ότι εγκρίθηκε, αλλά να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά ίσως. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται για τον 235. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Με μία ψήφο διαφορά απορρίπτεται. 237 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 238 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 239 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 240 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας Ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς 240. Άρχεται η ψηφοφορία για την 240. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ. Κατά αποχές Α ψηφίσουμε ηλεκτρονικώ, γιατί μπορεί να έχει μια ψήφο διαφορά. Προσπαθούμε λοιπόν να το επαληθεύσουμε γιατί 241. Άρχεται η ψηφοφορία, Πέρα. Με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. 242 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεν σηκώνω τα χέρια. 242. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε. Πέρας. Εγκρίνεται. 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 255 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 258 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 259 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 260 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 262 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 264 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 265 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έλεγχος, να ελέγξουμε για τη 265. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας με μία ψήφο διαφορά εγκρίνεται. 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14, 15, καταπίπτουν. 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ετυλογικές σκέψεις. 19, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20, υπέρ, κατά, αποχέ. Απορρίπτεται. 21. Έλεγχο, έλεγχο για την τροπολογία 20. 20. Θεολογική σκέψη. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν Πέρας. Με μία ψήφο διαφορά απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 μάλλον 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 με συγχωρείτε 29 πιπτή, 32 λοιπόν. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας επαληθεύσουμε. 36, Πίπερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο. Κάποιο ζήτησε έλεγχο. 39 λοιπόν. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. πέρα, Απορρίφθηκε. Σαράντα πέντε. Υπέρ. Σαράντα πέντε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ας κάνουμε έλεγχο. Όχι. Ωραία. Σαράντα έξι Υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε έλεγχο για τη 46. Όχι. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Όταν ε, θέλετε έλεγχο, δεν μπορείτε να φωνάζετε από πίσω, από το βάθος, τσεκ-τσεκ. Κάποιο να το ζητήσει σηκώνοντα το χέρι. Θέλει κανεί ε, επαλήθευση, κύριε Μπουτικόφερ. Ωραία. Επαλήθευση για την 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Με ισοψηφία απορρίπτεται. Ήταν σκόπιμο να ελέγξουμε, όντως. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση. Δεν θα συγχαρώ τον εισηγητή. Δεν θα ήταν σκόπιμο. Ταμείο συνοχής τώρα. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 και 12. 15 και 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η 16η τροπολογία. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3, 18 και 19 είναι πανομοιότυπες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται.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 Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 31. Λάμπερτ. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Η τροπολογία εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψεις 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση. Vous pouvez contrôler ici, hein? C'est Passiamo, sì, sì, come mm. controllo già il Eh, Je préfère eh, travailler sur le mio. Eh, passiamo al voto del ehm, provvedimento sugli strumenti. Καινοτόμο χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο του επόμενου πολιτής δημοσιονομικού πλαισίου. Καντσάν. Κομπρομέσο 1. Πρώτη τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 3. Τούρμς. Τούρμες. Εάν δεν σηκώνετε τα χέρια, δεν καταλαβαίνω. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Συμβιβαστική 2. Με συγχωρείτε. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχεδρίνεται. Συμβεβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 12, 12 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30. Δεν ψηφίζουμε την 29. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. 35. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον συνάδελφο Καντσιάνου. Επόμενο θέμα. Κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μαρτσίνκεβιτς. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Από... Με συγχωρείτε. Η ίδια ομάδα ψήφισε με διαφορετικούς τρόπου. Λοιπόν, τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Νομίζω ότι απορρίφθηκε, αλλά θέλω να το επαληθεύσω. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ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 Παρακαλώ εκείνοι που κάνουν τόσο θόρυβο στο βάθο να κάνουν λίγη ησυχία. Είναι ήδη περίπλοκη η δουλειά μα. Δεν χρειάζεται όλο αυτό ο θόρυβο. Λοιπόν, 19 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Έλεγχο για την τροπολογία 20 τη συναδέλφου Βερζά. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν πάντες πέρας. Εγκρίνεται. Με μικρή διαφορά, αλλά εγκρίθηκε. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική, άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Τελευταία συμφορία για σήμερα. δημιουργεί ενό μηχανισμού εταιρική σχέση με τη συνεργασία με τι τρίτε χώρε τη κυρία Τζαβέλα. Αρχίζουμε με την τροπολογία 19. Υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 20. Υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 6. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 21 η ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία εψήφισαν άπαντες πέρας απορρίπτεται Εάν μου επιτρέπετε μετά τα αυτήν την μακρά ψηφοφορία, μου έδωσαν λάθο πληροφόρηση από το γραφείο μου για την ψηφοφορία που πώ θα ψηφίσει το ΕΛΚ. Τέλο πάντων, απορρίφθηκε. 22. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε 9 της εισηγήτριας άρχεται η ψηφοφορία εξήφισαν άπαντες πέρας εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Με συγχωρείτε, 13 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε. 15 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται συγγνώμη 10... Ε, τροπολογία 17 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 καταπίπτει 5 υπέρ τα αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Έκθεση. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας για αυτή τη μακροσκελέστατη ψηφοφορία. Δύο λεπτά μόνον για Α συνεχίσουμε με την έκθεση του συναδέλφου Ρούμπικ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την ανταγωνιστικότητά τους και τις εμπορικές τους προοπτικές. Θα πρέπει όμως να περιοριστούμε λίγο γιατί είχαμε προβλέψει 45 λεπτά και έχουμε τελικώς μόνο 35. Συνάδελφε Ρούμπικ. Yeah, Το θέμα είναι σημαντικό. Έγιναν την Κυριακή οι εκλογές στην Ελλάδα. Για το μέλλον βέβαια η συνταγή δεν μπορεί να είναι περισσότερα χρέη και περισσότεροι φόροι διότι τότε θα γίνουμε ακόμα λιγότερο ανταγωνιστικοί στις εξαγωγές μας άρα θα προκύψει ακόμη μεγαλύτερη ανεργία. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε προϊόντα και εξαγωγές να μπορούν να προσφέρονται από εμά δηλαδή στη διεθνή παγκόσμια αγορά που να μπορούν να τα αγοράσουν και να θέλουν να τα αγοράσουν οι άλλοι καταναλωτές. Γι' αυτό και η ταξινόμηση αφενός διεθνοποίηση δηλαδή μείωση τη γραφειοκρατίας από την άλλη και επομένως τόνωση τη ανταγωνιστικότητα. Αυτά έχουν κέρια σημασία. Και ευχαριστώ ιδιαίτερως και τους συνεισηγητές και συνεισηγήτριες για τις συμβιβαστικέ τροπολογίες που έχουν κατατεθεί και νομίζω ότι όντως κάναμε μεγάλη πρόοδο και στα θέματα αυτά έχουμε επιτύχει ε, σημαντικό βαθμό συνένεσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω για την ώρα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν τώρα οι σκιώδεις ηγητές. Ε, είναι καταρχήν παρόν ο πρώτος και ο δισηγητής. Γιώχανσον. Παρακαλώ, κύριε Γιώχανσον. Sorry. Ε, Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, ήμουν αφηρημένος. Δεν φανταζόμουν ότι ήταν τόσο σύντομη η παρουσίαση του κυρίου Ρούμπιχ. Καταρχήν να τον ευχαριστήσω θερμά για την αγαστή συνεργασία που είχαμε. Ήταν πολύ επικοδομητικές συναντήσεις και οι συζητήσεις μας και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλο και μεγαλύτερη δέσμευση σε διεθνές επίπεδο και στη διεθνή αγορά και το εμπόριο υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι θεμελιώδου σημασία. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή προκειμένου να καταλήξουμε σε καλή συμφωνία και να αρθούν και οι φραγμοί που δημιουργεί η γραφειοκρατία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήταν πολύ επικοδομητική, επαναλαμβάνω, η συζήτηση και ευελπιστώ ότι θα καταλήξουμε και σε καλές συμβαστικές προτάσεις. Είναι σημαντικό να ε, ελαφρυνθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το γραφειοκρατικό άχθος, το διοικητικό άχθος γενικώ, αλλά το σημαντικό είναι να βρούμε μια λύση που θα ισχύει όχι μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και για τις υπόλοιπες, για να ενταχθούν ε, σε ένα γενικότερο πλαίσιο και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μην επιβάλλεται επιπλέον διοικητικό άχθος σε αυτές. Πάντως, επαναλαμβάνω, ήταν ε, πολύ καρποφόρα η συνεργασία μας με τον εισηγητή, τον κύριο Ρομπίχη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπιτικόφερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομος. Συμφωνώ με τον συνάδελφό μου Γιώχανσον και μόνο για το θέμα της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης θέλω να αναφέρω κάτι το συγκεκριμένο. Το έχουμε συζητήσει και εκτός σκιωδών εισηγητών. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό. Εμένα θα μου άρεσε η high level group η οποία ασχολείται ήδη, υπάρχει και ασχολείται ήδη με το θέμα να την βάλουμε αυτήν στο τιμόνι και να πούμε ότι το Κοινοβούλιο θα ήθελε αυτή η ομάδα υψηλού επίπεδου να κάνει προτάσεις και στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο και μάλιστα τακτικά να υποβάλει μάλιστα ευθέως τις προτάσεις αυτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς να αναλάβουμε δράση στην βάση αυτών των προτάσεων. Αυτό θα είναι πολύ πιο στοχευμένο, διότι αυτή η High Level Group διαθέτει και την εμπειρογνωμοσύνη. Καλύτερα έτσι παρά να βάλουμε ποσοτικούς στόχους για την μείωση της γραφειοκρατίας. Νομίζω ότι αυτή η ιδέα μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικοδομητική. Η κυρία Φόρντ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την συνεργασία. Κοιτάξτε τι γίνεται με την ευρωπαϊκή οικονομία και ειδικά με τις μικρές επιχειρήσεις. Αντιμετωπίζουν μια κρίση εμπιστοσύνης. Ε, μάλλον οι ίδιες δηλαδή βρίσκονται σε μια κρίση εμπιστοσύνης. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει καλύτερο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό εμείς ως πολιτικοί γυναίκες και άνδρες να συμπαραταχθούμε μαζί τους και να το δηλώσουμε αυτό σαφώς, να δουν δηλαδή ότι εμείς νοιαζόμαστε και προσπαθούμε. Όλοι λέμε ότι θέλουμε να μειώσουμε το επίπεδο της γραφειοκρατίας και να την περικόψουμε. Και βέβαια θέλω να τους το δηλώσουμε αυτό καθαρά, να μπορούμε να τους πούμε ότι οι μικρές επιχειρήσεις είναι αθώες μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου, ότι θα τις βγάλουμε απ' έξω από τις νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι ότου αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητο να υπάρξουν κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις και να ενταχθούν σε κάποια νομοθεσία. Αυτό θα είναι ένα μήνυμα εμπιστοσύνης προς τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε βεβαίως να κάνουμε μια κοινωνία δύο επιπέδων. Έχει δίκιο ο κ. Γιώχανσον. Αλλά όπου δεν χρειάζεται να ρυθμίσουμε, δηλαδή στο τμήμα εκείνο της ε, αλυσίδας της προσφοράς όπου δεν χρειάζεται, να τους το πούμε αυτό καθαρά, να κάνουμε καθαρά τη δήλωση ότι αυτή ότι είμαστε στο πλευρό τους, ότι θέλουμε να ισχύουν καθεστώτα ελαφρά, να μην επιβαρύνονται οι μικρές επιχειρήσεις. Το άλλο θέμα το οποίο συχνά μου τίθεται υπόψη δεν είναι μόνο των τραπεζικών δανείων, αλλά και άλλες τραπεζικές και άλλων τραπεζικών υπηρεσιών και κυρίως για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες ε, έχουν και ε, συναλλαγματικές υποθέσεις, δηλαδή χρησιμοποιούν διαφορετικά νομίσματα. Μιλώντας με τις επιχειρήσεις αυτές βλέπουμε συχνά πρώτα-πρώτα πόσο καιρό χρειάζεται για να ε, εκαθαριστεί μια επιταγή, αν θα είναι σε δολάρια ή σε άλλο νόμισμα μπορεί να μετατραπεί εύκολα από το ένα νόμισμα στο άλλο, να πληρωθεί σε άλλο νόμισμα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε επιγόντως να εξετάσουμε τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες υπέρ των μικρών επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, όπου για παράδειγμα ίσως η νομοθεσία για το ξέπλυμα του χρήματος περιπλέκει τα πράγματα περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο για να συλλαμβάνονται οι κακοί, οι εγκληματίες δηλαδή. Ένα παράδειγμα, χρειάστηκε μια μικρή επιχείρηση έξι μήνες για να εισπράξει μια επιταγή της IBM. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Μάλιστα. Θα ήθελα να μιλήσω και εγώ εν συντομία ως και όδη συγκήτρια της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο Ρούμπικ για την ε, πολύ ευρυθή του ε, έκθεση και νομίζω ότι ήταν πολύ αξιόλογη. Όλοι καταθέσαμε τροπολογίες, δεν θα επιμείνω στα επιμέρους Πιστεύω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, περιμένουν συγκεκριμένες προτάσεις και όχι άλλη κολυσιεργία. Θέλουμε να ε, ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκώντας τις αρμοδιότητές της να υθετήσει συγκεκριμένα μέτρα για θέματα που έχουμε διευκρινίσει, γιατί γνωρίζουμε ποια είναι τα δεινά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπερβολική γραφειοκρατία, δύσκολη πρόσβαση στο δανεισμό είτε και είστε στα τραπεζικά δάνεια, αλλά και στην οργάνωση των τραπεζικών υπηρεσιών. Και επίση έχουν κάποιε δυσκολίε και με, και με τη δημόσια διοίκηση και απέναντι στι μεγάλε επιχειρήσει. Θα πρέπει να έχουν και με τη δημόσια διοίκηση και με τι άλλε επιχειρήσει, σχέσει που δεν θα τους δημιουργούν προβλήματα. Πιστεύω ότι ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε και με την ομάδα Υψηλοπέδου συμφωνώ με τον κύριο Μπουτικόφερ και ήδη ο κύριος Ρούμπιχ στην έκθεση του έχει πολλές προτάσεις, θα καταθέσουμε και εμείς κάποιες τροπολογίες, να ασχοληθούμε και με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πραγματικά σημαντική κληρονομιά της ευρωπαϊκής οικονομίας έχουμε εργοδότες που συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις τους, αλλά έχουμε και εργαζόμενους που αισθάνονται ότι είναι τμήμα αυτών των επιχειρήσεων, ότι ανήκουν σε αυτή την επιχείρηση και θέλουμε μία αρμονική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των, εργαζομένων, των σχέσεων των εργαζομένων και των εργοδοτών, ώστε με στενή συνεργασία και αρμονική συνύπαρξη να ενισχυθεί η θέση των επιχειρήσεων. Γιατί σε ορισμένες επιχειρήσεις η μικρή διάσταση δεν εγγυάται σε τελική ανάλυση και κάποια θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Θα πρέπει λοιπόν και τα δικαιώματα των εργαζομένων να τα λάβουμε υπόψη και θα ήθελα ο εισηγητή να διευρύνει κάπως την εκθέση του ώστε να συμπεριλάβει και αυτά τα θέματα και τι πτυχέ των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Έτσι θα ενισχύσουμε και δεν θα επιβαρύνουμε τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, γιατί οι σοβαροί εργοδότες αυτό μα λένε ότι η, η επιτυχία του οφείλεται και στη δική του προσωπική ανάπτυξη αλλά και στην ενεργό ανάμειξη και το ζήλο και των εργαζομένων του. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Ρούμπιχ για την πολύ αυτή σημαντική του έκθεση. Και αν δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ζουλιάν Γκεργέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ευαρέσκειά τη για την σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή Βιομηχανία Έρευνα και Ενέργεια για την έκθεση του κυρίου Ρουμπίχ. Όπως είπαμε και κατά την αρχική παρουσίαση της έκθεσης, ε, φαίνεται μια σαφής δέσμευση και στράτευση υπέρ των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλη ε, υποστήριξη της, ε, των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευφυή e ρύθμιση και την ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο γενικότερο πλαίσιο, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση. Σε ό,τι αφορά τις προτινόμενες τροπολογίες θα ήθελα να κάνω δύο διευκρινήσεις. Η πρώτη αφορά την διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες δράσεις που προτείνονται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα υποβληθούν μέχρι τα τέλη του 2012, προβλέπονται πολλά μέτρα. Καταρχήν μια απογραφή των υφιστάμενων μέτρων στα κράτη-μέλη. Κατόπιν, ένα εντοπισμό των κενών και των αδυναμιών, δηλαδή των ε, υπηρεσιών που δεν ε, υπάρχουν για να στηρίξουν την αλλοδαπή της μικρομεσαίας μας επιχειρήσεις. Και επίσης το 2013 θα γίνει μετά από αυτή την απογραφή και την ε, επισκόπηση μία άντληση συμπερασμάτων για να δούμε τι συστάσεις θα υποβάλουμε και τι μέτρα χρειάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να, να γίνει ένας ε, απολογισμός, ένας κατάλογος των μέτρων και όχι φυσικά μία αποδυνάμωση των υπηρεσιών ε, που προσφέρονται ήδη από τα κράτη-μέλη, όπως φαίνεται να υποδεικνύουν μερικές πρωτοβουλίες. Ό,τι αφορά το δίκτυο των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Όπως δείχνουν οι τροπολογίες, πολλές τροπολογίες, θα πρέπει να ενισχύσουμε την ορατότητα, την αποτελεσματικότητα και την διακυβέρνηση αυτού του δικτύου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Συμφωνούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θέλουμε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Και μάλιστα οι εταίροι των δικτύων ε, επιλέξαν μετά από διαγωνισμό και μάλιστα θα προκηρυχθεί νέα πρόταση για υποβολή προσφορών. Ελπίζουμε να λάβουμε μέσω του νέου αυτού διαγωνισμού τα καλύτερα προγράμματα και σχέδια. Έχουμε επαφέ και με τι διαφορέ οργανώσει ε, επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ετοιμάσουμε μια νέα δομή διακυβέρνηση για αυτό το δίκτυο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει πάλι ο συγκεκριτή ο κ. Ρουμπίχ για να δευτερολογήσει. Ελπίζουμε να είναι και στη δευτερολογία του εξωσύντομο όσο στην αρχική του παρατήρηση. Θέλω μόνο να ευχαριστήσω τις και, τις και τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο κάνει μαζί με την Κομισιόν ένα σημαντικό βήμα προς ένα σταθερότερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Και όπως ξέρετε η ψηφοφορία θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου είτε στην επόμενη συνεδρία στις 17 με 18 Σεπτεμβρίου ανάλογα με την πορεία των εργασιών μας. Επόμενο σημείο, οι κανόνες ε, και δια... Ε, συμμετοχής και διάδοση του προγράμματος πλαίσιο έρευνας και καινοτομία ορίζον 2020. Κανόνες διάδοση των αποτελεσμάτων. Το λόγο έχει ο ο κύριος Κρίστιαν Έλερ. Κυρία Πρόεδρε, φοβούμαι ότι δεν θα μπορώ να είμαι τόσο σύντομος όσο ο κύριος Ρούμπικ. Θα προσπαθήσω πάλι στα αγγλικά. Θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τους άλλους σκιώδεις ηγητές και αυτό δεν το λέω τυπικά. Το Κοινοβούλιο με τους κανόνες για το πακέτο για τον ορίζοντα το Κοινοβούλιο έρεται στο ύψος των περιστάσεων. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω το περιεχόμενο της εκθέσεώς μου. Θα προσπαθήσω μόνο να αναφερθώ σε ορισμένα σημαντικά θέματα. Ναι, πρόκειται για απλούστευση, αλλά και αποτελεσματικότητα για τη συμμετοχή της βιομηχανίας, για την μετακίνηση προς την καινοτομία ε, και για τον προϋπολογισμό του ορίζοντα 2020. Θα ήθελα πρώτα να πω ότι ε, συμφωνώ με τις προτάσεις της Κομισιόν για την απλούστευση, για αυτή την μετακίνηση προς ε, την καινοτομία και νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνουμε είναι προσπάθεια προσαρμογής όχι όμως μόνο πολιτικού ή συμβολικού χαρακτήρα προς την κατεύθυνση μιας απλούστευσης, αλλά αυτό που επιδιώκουμε είναι να επιτύχουμε μια αποτελεσματικότητα, μια αποδοτικότητα. Το ερώτημα δηλαδή είναι πόσο αποδοτικό θα είναι το νέο αυτό πρόγραμμα. Η απλούστευση αποτελείται από τρεις πυλώνες. Πρώτα, ένα σύνολο ξεκάθαρων κανόνων για τις αρμοδιότητες με PPP, GTI κτλ. Και όλα αυτά σε ένα στόχο ορίζοντα 2020, άρα με μια καλύτερη διάρθρωση και συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους ε, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Επίσης για τις, ε, πρακτικές, τις λογιστικές πρακτικές προς όφελος των συμμετεχόντων που θα καταλήξουν και στους δημοσιονομικούς κανονισμούς έτσι ώστε να ληφθούν περισσότερο υπόψη οι πρακτικές των χωρών μελών. Ένα σύστημα ποσοστών επιστροφών που θα λαμβάνει υπόψη το πλήρες κόστος και που θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις διαφορετικές χρηματοδοτικές ανάγκες των διαφόρων συμμετεχόντων και η πρότασή μας ίσως να κάνει το, την όλη προσέγγιση πιο αποτελεσματική για τους συμμετέχοντες. Δεν πρόκειται για καμιά υπεραπλούστευση. Το κείμενό μου είναι πάρα πολύ πολιτικό. Είναι σχετικά περιορισμένο σε μήκο. Βέβαια και μέσω τη διακλαδική διαπραγμάτευση να προκύψει από αυτό, αλλά χρειάζεται να βλάβει και περισσότερο πρακτικό χαρακτήρα. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα λογικό βήμα προ τα Εμπρό. συνέχεια όπου αυτό είναι αναγκαίο και το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι, με full cost option, Δεν έχει νόημα δηλαδή να εξαναγκαστεί κάποιος να κινηθεί προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Διαφορές του επίπεδου χρηματοδότησης για τους διάφορους ενδιαφερόμενους, όπως έχουμε συμφωνήσει για παράδειγμα για τη σημασία των μικρών και μεσών επιχειρήσεων, να έχουμε σημαντική έντονη συμμετοχή των μικρών και μεσών επιχειρήσεων με προβολή του δικού τους ενδιαφέροντος και συμφέροντος. Επίσης, μείωση των δραστηριοτήτων και των funding rates και λήψη υπόψη των λογιστικών πρακτικών των χωρών μελών. Δεύτερο, πώς θα συμμετάσχουν οι κράτη περισσότερο στο πρόγραμμα. Πιστεύω και πρέπει να δούμε τα πράγματα ρεαλιστικά ότι η αύξηση της χρηματοδότησης που προτείνει για τις συμμετέχουσες βιομηχανίες η Κομισιόν έχει άμεση σχέση με το ποιο προπολογισμό έχουμε στη διάθεσή μα. Με δεδομένο τον προπολογισμό, με μια αύξηση της τάξης του 6% περίπου, είναι βέβαια ενδιαφέρον, αλλά πώς θα γίνει να προσελκύσουμε τους ενδιαφερόμενους κλάδους με υψηλότερα ποσοστά χρηματοδότησης αλλά πώς θα συμμετάσχουν σε ένα άκαμπτο πρόγραμμα ή θα μπουν μόνο επειδή θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Αύξηση λοιπόν της ε, συμμετοχής ε, της βιομηχανίας, αλλά τελικά με υψηλότερα ποσοστά. Αναλογικά δηλαδή. Άρα θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή της βιομηχανίας, αλλά όχι τόσο σε αριθμούς μονάδων, αλλά περισσότερο σε χρηματοδότηση ποτέ δεν έχουν παραπονεθεί ότι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 2 ήταν πολύ χαμηλό. Έχουν παραπονεθεί για το ότι η διοικητική επιβάρυνση και η λογιστική επιβάρυνση ήταν πολύ υψηλέ. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς έχουμε προσπαθήσει να ανταποκριθεί σε πολλές από τις ανησυχίες αυτές, να ανταποκριθούμε σε πολλές από τις ανησυχίες αυτές. Το όριό μας είναι κατά μέγιστον όρων 6 μηνών και αν δούμε ότι σε σχέση με τα διεθνή benchmark, ακόμα και αν τα καταφέρουμε μέσα σε έξι μήνες, δεν θα έχουμε προχωρήσει αρκετά. Θα βρισκόμαστε κάπου στο μέσον. σε ό,τι αφορά τη σύγκρισή μας με το διεθνές περιβάλλον. Η συμπερίληψη της full cost option είναι υπέρ της βιομηχανίας και βέβαια η χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι σημαντικό και για να συνδυάσουμε τον ορίζοντα 2020 και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Για παράδειγμα τα ε, διαφθορτικά ταμεία αλλά και άλλες πηγές. Με ξεκάθαρους κανόνες για ανοιχτή πρόσβαση και IPR αυτά όμως υπό την προϋπόθεση ότι θα βρούμε μια ισορροπία της πρόσβασης και της βιομηχανίας και βέβαια για τα GTI και άλλα PPP. Δυστυχώς ο Αγγλωτής χρησιμοποιεί πάρα, πολλές, πάρα πολλά ακρόνημα χωρίς να εξηγεί περί τίνος πρόκειται. Η συζήτηση στο Συμβούλιο με ανησυχεί. Χθε συναντήθηκα με εκπροσώπους μιας μεγάλης ευρωπαϊκής χώρας και φαίνεται όμως ότι προβλέπουν σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό. Και εδώ τίθεται το θέμα των ποσοστών παρεμβάσεων. Ήδη η Κομισιόν προβλέπει τις τάξεις του 7% τώρα αυξήσει τη τάξη του 7%. Αν όμως τελικά αποδειχθεί ότι θα έχουμε λιγότερα χρήματα στη διάθεσή μας, θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τη μόχλευση. Η αύξηση του αποτελέσματος μόχλευσης στον ορίζοντα 2020 θα έχει θετική επίπτωση στις χρηματοδοτήσεις έρευνας και ανάπτυξης. Όχι να δώσουμε περισσότερα λεφτά σε λιγότερους, αλλά να βρεθεί μια ισορροπία στην μόχλευση μεταξύ έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας και όπως είπα η προσέγγιση μας πρέπει να είναι ρεαλιστική μέσα σε ένα περιβάλλον όπου ίσως έχουμε μια αύξηση της τάξης του 6%. Αυτό βέβαια πρέπει να οδηγήσει σε μια πολύ προσεκτική συζήτηση για τα ποσοστά παρεμβάσεων. Ευχαριστούμε τον κύριο Έλερ. Ξεκινάμε με τους κοιόδης εισηγητές. Ο κύριος Γκλάντε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ας φέρω ένα παράδειγμα από τη φυσική. Μιλούμε εδώ για ένα σύστημα κινήτρων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κάποιες προτάσεις απλουστεύσεων Καμιά φορά όμως οι δονήσεις είναι υπερβολικά υψηλές. Δηλαδή η Κομισιόν έχει προχωρήσει σε μια υπεραπλούστευση. Ο κύριος Έλερ με την πρότασή του, με τις προτάσεις του, ε, τα περιπλέκει κάπως τα πράγματα. Πρέπει να βρούμε ένα μεσαίο δρόμο. Αυτό που θέλουμε είναι οι κανόνες να είναι ευκολότεροι, η συμμετοχή να είναι επίσης ευχαιρέστερη. Μπορούμε να μιλήσουμε βέβαια για τα ποσοστά επιστροφών για τη συμμετοχή. Στα πλαίσια του 7ου προγράμματος, ε, του 7ου προγράμματος είχαμε τις ρυθμίσεις για τις ποσοστώσεις επιστροφές για τα πανεπιστήμια για παράδειγμα. Εκεί πρέπει να βρούμε ένα υγιή συμβασμό. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι, αυτό το είδα και στις συζητήσεις που έχω διεξαγάγει και μου υποβλήθηκε, είναι οι πολύ, διαφορετικές, τα, πολύ διαφορετικοί τρόποι υπολογισμού για το κόστος προσωπικού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εάν απασχολώ λοιπόν μια ε, Βελγίδα συνεργάτηδα με το βελγικό δίκαιο ω βάση είναι πολύ διαφορετικό από ότι έχω μια, έχω μια Γερμανίδα με το γερμανικό δίκαιο. τα συστήματα αυτά πρέπει να αναγνωριστούν και πρέπει να διασυνδεθούν το, τα εθνικά. Τώρα, το time to grant, δε, μέχρι ότου δηλαδή ένα ε, πρόγραμμα λάβει τη χρηματοδότηση. Οι έξι μήνες είναι φιλόδοξος στόχος, χωρίς βέβαια να υπάρξει κενό ώστε να γίνει πάλι καθυστέρηση, δηλαδή να αναβληθεί η εφαρμογή του έργου διότι λείπουν κάποια έγγραφα κτλ. Επαναλαμβάνω, το εξάμεινο είναι φιλόδοξο στόχος. Τρίτο, το 7% ε, κόστο διαχείρισης, management. Βέβαια, το management μια κοινοπραξία δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά 7% μου φαίνεται ότι είναι πολλά λεφτά που χάνει βεβαίω η έρευνα. Πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν αν όντω αυτό το επίπεδο του 7% είναι αιτιολογημένο ή μήπως πρέπει να μειωθεί. Τέταρτο σχόλιο, όπως είπε και άλλος συναδελφός προηγουμένως, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Πού βρίσκεται η μηπως πρεπει να μειωθει τεταρτο σχολιο οπως ειπε και άλλο συναδελφο προηγουμένω, δικαιωματα βιομηχανικης ιδιοκτησία που βρισκεται η ισορροπια μεταξυ του open access και το όριο όπου θα πούν οι βιομηχανίε. «Α, αυτό μα φαίνεται πολύ επικίνδυνο, δεν συμμετέχουμε». Αυτά λοιπόν για μένα είναι τα πιο θεμελιώδη θέματα. Το άλλο είναι ε, τα κέντρα αριστείας που τα έχουμε ξανασυζητήσει. Εδώ πρέπει να επανείδουμε τον ε, ορισμό. Κάποιος ασυνάδελφος θεωρεί ότι εκεί χάνονται κάποια ε, κονδύλια. Για να επιτύχουμε την αριστεία, το έχουμε δει και από το παρελθόν, πρέπει να δημιουργηθεί μια υποδομή. Εκεί όμως δεν είναι η σωστή επιλογή η πηγή του ταμείου αυτού. Έχουμε λοιπόν ακόμα δουλειά μπροστά μας. Η συνεργασία όμως λειτουργεί καλά. Και μετά από τις θερινές διακοπές νομίζω θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αρκετά ταχύ ρυθμό. Άλλωστε μετά από τις θερινές διακοπές θα γνωρίζουμε και ε, πιο, ποια κονδύλια θα διαθέτουμε και δεν θα είμαστε μονάχα στο 6%. Ο κύριος Γιώχανσον. Thank uh, also... Ευχαριστώ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή μας, τον κύριο Έλερ, γιατί όπως είπα και χθες στους υπόλοιπους και ηγητές ήταν πολύ σημαντική συζήτηση και έμπνευση και για τον ορίζοντα 2020. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ποσοστό συμμετοχής, χαίρομαι που το περιλαμβάνουμε εδώ και ο κύριος Ελερίδη από την αρχή είπε ότι ο διάβολος κρύβεται μέσα στις λεπτομέρειες. Αλλά μερικές φορές και οι ήρωες φαίνονται στις λεπτομέρειες. Φυσικά θα πρέπει να συζητήσουμε και τα πολιτικά μηνύματα, αλλά αν μπορούμε να βρούμε καλούς κανόνες συμμετοχής, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική η φιλοδοξία του κυρίου Έλερ για γενική απλούστευση και ε, επίτευξη ενός ενιαίου ε, πακέτου κανόνων. Θέλουμε ένα ευρύτερο φάσμα περισσότερων δραστηριοτήτων και περισσότερων συμμετεχόντων που θα καλύπτονται από τους νέους κανόνες χρηματοδότηση. Γιατί όπω είπαμε έχουμε διαφορετικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρξει μια μεγαλύτερη ομοιομορφία. Σε ό,τι αφορά τα ποσοστά χρηματοδότηση, σε σχέση με το ερευνητικό πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο 7, υπάρχει κάποια βελτίωση, αλλά σε σύγκριση με τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε νέε περιπλοκέ που θα ε, αυξήσουν ε, άσκοπα το γραφειοκρατικό άκθο. Όπω είπα όμω και στη συνεδρία των σχεδόν εισηγητών, έχουμε ένα πολύ καλό σημείο εφετηρία. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση και ίσω εμεί θα αναδειχθούμε ε, ω οι ήρωες των λεπτομεριών. Είμαι υπέρ μια μεγαλύτερη αποδοχής ε, των συνήθων λογιστικών πρακτικών και των δικαιούχων. Είναι σημαντικό μήνυμα της απλούστευσης που επιζητούμε. Σε ό,τι αφορά τις διάφορες ε, τιμές, ιδιαίτερα το inducement price. Είναι πολύ καλό ε, σημαντικό και συμπληρωματικό μοντέλο που είχαμε υποστηρίξει στην ομάδα και χαίρομαι που κύριε Έλερ το περιλάβατε αυτό στην έκθεσή σας. Ε, θα, επίσης είμαι υπέρ της βράξης της προθεσμίας εξάμεινο για τις επιχορηγήσεις, ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι και εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε διαφορετικούς μηχανισμούς ώστε να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν συνεχή ενημέρωση για το σε ποια φάση της ε, έγκρισης βρίσκονται. Μιλήσαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, είμαι υπέρ των, ε, της μεγαλύτερης ανάμειξης ενσωμάτωσης τους στο πλαίσιο αυτό, αλλά να μην ξεχνούμε και το θέμα της ισότητας των δύο φύλων θα πρέπει στους κανόνες της συμμετοχής να έχουμε υπόψη και τη διάσταση της ισότητας των φύλων. Γιατί εκεί βρίσκεται η ισχύ της Ευρώπης, ε, στην ε, γενικευμένη συμμετοχή, να μπορούν όλοι να λαμβάνουν μέρος. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε την προσπάθειά μας για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών. Νομίζω ότι στα πλαίσια τη συζήτηση για του κανόνε συμμετοχή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη διάσταση του φύλου. Ευχαριστώ. Grazie, la parola alla collega Ford. Ευχαριστούμε κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Κρίστινα για την πολύ και σκληρή δουλειά που έκανε για, τις, για το ποσοστά χρηματοδότηση και τη σχετική κατάσταση. Για το ζήτημα λοιπόν αυτό εγώ δεν έχω ακούσει επιστήμονε και επιχειρήσει να μου λένε ότι θέλω να συμμετάσχω σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, εάν το ποσοστό είναι τόσο ή τόσο. Όχι, ειδικά οι μικρέ επιχειρήσει μου λένε δεν θέλω πλέον να συμμετέχω, γιατί η γραφειοκρατία είναι πάρα πολύ και τα έντυπα πρέπει να συμπληρώσει κανεί ε, πάρα πολλά και χρειάζονται και πάρα πολλοί μήνε μέχρι να λάβω το οποιοδήποτε ποσό. Λοιπόν, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει η απαραίτητη μόχλευση με άλλη χρηματοδότηση διότι δεν υπάρχουν πλέον δημοσία κονδύλια. Νομίζω ότι η προσέγγιση του Κρίστια να προσπαθεί να εξεύει διαφορετικού τρόπου, να υπάρξει μόχλευση από διαφορετικού τομεί και εξυπηρετική είναι και διευκολύνει τα πράγματα. Και εγώ έκανα μια τροπολογία σε σχέση με τα ποσοστά, αλλά νομίζω ότι καλώ τα πρότεινα όπω τα πρότεινα. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ότι σε διαφορετικού τομεί ε, τη επιστήμη χρειάζεται και διαφορετική χρηματοδότηση από διαφορετικού τομεί. Δηλαδή μια εταιρεία ε, IT που μπορεί να αναπτύσσει μια εφαρμογή για το iPhone πριν από το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα έπρεπε να λειτουργεί διαφορετικά από κάποιους άλλους που μπορεί να αναπτύσσουν φάρμακα ή βιοτεχνολογικά προϊόντα και να χρειάζονται και δεκαετία. Είναι λοιπόν διαφορετικά, διαφορετικές ανάγκες του κάθε επιστημονικού κλάδου. Επίσης, συμφωνώ με την μέθοδό σας για τον υπολογισμό του πλήρους κόστους. Αυτό μπορεί να διευκολύνει σε κάποιες Τώρα για να πλουστεύσουμε τα γραφειοκρατική διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει ένας κώδικα πρακτικών όπου να προβλέπονται και κάποια στοιχεία από την πράξη για τι μικρέ επιχειρήσει, λόγω χάρη στι σχέσει που θα πρέπει να έχει κανεί με τι μικρότερε επιχειρήσει και του συμμετέχοντε. Για τον ε, χρόνο τη ε, απονομή των ε, βοηθειών, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι Μόλις την περασμένη εβδομάδα περισσότεροι πήραν την έκθεση αυτής της ε, γλώσσες τους και πρέπει να υποβάλουν τροπολογίες μέχρι την επόμενη Τρίτη. Ε, αυτή είναι μια από τις ανατροπές που δεν θέλουμε να έχουμε, μια από τις δυσκολίες που δεν θέλουμε να. στι οποίε δεν θέλουμε να υποβάλουμε τι μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει να υπάρχει ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να λαμβάνει υπόψη και τις ε, διακοπές ενδεχομένως των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ή άλλους επιχειρηματικούς κύκλους. Στα σχόλια που είδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση των 12 για την ε, διαδικασία αιτήσεων σε δύο στάδια, αυτό σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι εύστοχο σε ορισμένου διαγωνισμού. Τέτοιου είδου ευελιξία όμως δεν θα πρέπει να περιπλέκει περαιτέρω τα πράγματα ίσως να απλουστεύσει σε ορισμένες περιπτώσεις την κατάσταση. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό, βελτιώσεις και στη διαφάνεια χρειάζεται και καθώς και εμπιστοσύνη στη διαδικασία της ε, διόρθωσης, της επίλυσης διαφορών. για την επιστροφή δαπανών. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να δούμε κατά πόσον περισσότερα σχόλια μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινή διακοπή για να τι καλύψουμε και στι τροπολογίε. Ο Λάμπερτ είναι ο τελευταίο και ο αν θέλετε, και μετά θα δούμε του υπόλοιπου ομιλητέ. Δεν θα σχολιάσω φυσικά όλα α, τα σχόλια του Κρίστιαν, γιατί συμφωνώ με πολλές από τις παρατηρήσεις του και καλό είναι να τονίζουμε και τα κοινά μας σημεία, όχι μόνο τις διαφωνίες. Σε ό,τι αφορά τη μόχλευση, ακούσαμε πολλές φορές τη λέξη μόχλευση στην ομιλία του Κρίστιαν και όπως είπα και χθε είναι κάτι που φαίνεται ότι μας έχει γίνει έμονη ιδέα αυτή η μόχλευση. Θέλουμε τα δημόσια κονδύλια, τα κρατικά κονδύλια και οι κρατικές επενδύσεις να, γίνουν, να δημιουργούν μόχλευση για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Και βέβαια η όρεξη για τις ιδιωτικές επενδύσεις δεν είναι ίδια σε όλους τους τομείς, αλλά με ενοχλεί κάπως το γεγονός ότι ε, βλέπω πώς οι έμονοι έχουν μερικές φορές οι επιχειρήσεις με, τη, με το βραχυπρόθεσμο και όταν χρειάζονται μακροπρόθεσμες προσπάθειες και επενδύσεις φαίνεται ότι ε, δηλιάζουν οι επιχειρηματίες. Και έτσι ο δημόσιο φορέα, ο δημόσιο τομέα είναι τελικά ο μόνο που ασχολείται με τι μακροπρόθεσμε επενδύσει που ίσω είναι και πιο ρηψοκίνδυνε. Ενώ ο ιδιωτικό τομέα ουσιαστικά ντρέπει καρπού από πολύ βραχυπρόθεσμε προσπάθειε και επενδύσει. Διαφωνώ λοιπόν αυτή την προσέγγιση. Αν θέλουμε ο δημόσιο τομέα να επενδύει στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, ε, να μπορούν και οι ιδιώτες να επενδύουν σε τέτοια είδους σχέδια. Έτσι θα δημιουργηθεί μόχλευση από γενικευμένη συμμετοχή. Έτσι θα αυξηθεί το αποτέλεσμα της μόχλευσης με κοινή συμμετοχή σε μακροπρόθεσμα σχέδια και των ιδιωτών. Νομίζω ότι αυτό το μερίδιο της βιομηχανίας θα πρέπει να ενισχυθεί στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Επίσης, ο Κρίστιαν έκανε μια αρχικά απλή πρόταση πολύ πιο περίπλοκη μία ακόμη φορά, αλλά νομίζω ότι την έκανε και ξυπνότερη με τις επιπλοκές που εισήγαγε. Γιατί είδαμε την πρόταση των Πρασινών και εκεί ίσως τα ποσοστά χρηματοδότησης για δραστηριότητες κοντά στην αγορά ήταν υπερβολικά γενναιόδοροι. Και ίσως εκεί είναι η ε, εύκολη καρπή και το εύκολο κέρδος. Ε, γιατί είχαμε το 70% της ε, κοινοτικής χρηματοδότησης για το επιλέξιμο κόστος. Ο Κρίστιαν όμως φρόντισε να γίνει πιο σοφή, έξυπνη η πρόταση. Τώρα, για τη διάδοση και το ανοιχτή πρόσβαση, το open access, είναι μια ε, πράξη εξισορρόπηση, γιατί δεν είναι γιατί δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα. Υπάρχουν και διάμεσες λύσεις. Εμείς θα προτιμούσαμε την ανοιχτή γνώση, μάλλον και γνωρίζουμε ότι για να δημιουργηθεί καινοτομία θα πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερη γνώση. Βέβαια δεν είμαστε και αφελείς. Θέλουμε η καινοτομία να αποφέρει και καρπούς, να δημιουργεί και κέρδος. Δεν θέλουμε εμείς μόνο με τις επενδύσεις και άλλοι να καρπώνονται τα κέρδη και τα ωφέλη αυτών των επενδύσεων. Θέλουμε μια σωστή εξισορρόπηση. Κρίστιαν, προτείνει εδώ εξαίρεση των ε, χρηματοδοτήσεων από του κανόνε για, το, για τις κρατικές ενισχύσεις. Με προβλημάτισε αυτό. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρώπη είναι ένα άλλο επίπεδο διακυβέρνηση. Καταγόμαστε και δύο από ομόσπονδες ε, χώρε και νομίζω ότι Ομοσπονδιακέ χώρε, και νομίζω ότι το πλαίσιο της, ε, της δημόσιας και οι κανόνε κρατικών επενδύσεων ίσω δεν ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ίσω μάλλον παρεξήγηση υπάρχει εδώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφωνία επί της ουσίας. Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι αυτό το 7% κατά αποκοπή ποσό για το διοικητικό έχθος. Άχθος. Είναι πολύ απλή και άμεση αυτή η πρόταση. Το κόστος διαχείρισης δεν δημιουργεί κατά ανάγκη αύξηση του κόστους του σχεδίου. Υπάρχει και ένα πάγιο τμήμα και υπάρχει και ένα μεταβλητό τμήμα σε αυτό το κόστος. Εδώ δύο είναι οι λύσεις. Είτε θα πούμε ότι έχουμε ένα πάγιο διαχειριστικό κόστος που το αποζημιώνουμε ή έχουμε ένα φθήνοντα συντελεστή που μπορεί να είναι 7%, για τα μικρά, 7 για τα μικρά σχέδια, αλλά μετά θα μειώνεται, ε, θα γίνεται 6, 5, 4 για τα μεγαλύτερα σχέδια. Είμαι υπέρ της απλότητας. Δεν θέλουμε με υπερβολικές περιπλοκές ε, να καταπνίξουμε την προσπάθεια ή δεν θέλουμε υπερβολικές επιστροφές. Θέλουμε έναν απλό συντελεστή, αλλά να έχει φθήνοντα χαρακτήρα, να μειώνεται σταδιακά για να μην γίνεται υπερβολική επιστροφή του διοικητικού κόστους. Και τέλος, κάτι που αναφέρεται ακροθυγός και στο εξαπλό πακέτο, τα GTIs. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, Κρίστιαν, αλλά όσο περισσότερο μιλώ με εκπροσώπους της βιομηχανίας, όσο περισσότερο μιλώ με ακαδημαϊκούς, τόσο περισσότερο ακούω αρνητικά σχόλια για τα GTIs τις κοινέ τεχνολογικές ε, πρωτοβουλίες. Εγώ είμαι, ήμουν αρχικά υπέρ της διεύρυνσης. Κάπως μου είπε ότι το καλό με τα JTIs είναι ότι ε, η εμπειρία μας δίδαξε τι θα πρέπει να αποφύγουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αποφύγουμε. Αν εσείς ακούσετε ε, θετικά σχόλια για τα JTIs θα μου τα πείτε. Ίσως όχι εδώ, μπορούμε και διμερώς να τα εξετάσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Έλερ για τα θέματα της χρηματοδότησης, για τις απλουστεύσεις, αλλά ως εκπρόσωπος μιας χώρας που δυστυχώς ε, σε αυτό το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο ε, δεν κατάφερε να διευκολύνει τα ερευνητικά θέματα. Για παράδειγμα, στις αρχές της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας, όταν ξεκίνησε το έβδομο ε, πρόγραμμα, από τις 200 αιτήσει μόνο κάποιες δεκάδες έγιναν δεκτές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αφενός έχουμε ε, υπαλλήλου, ε, χρήματα, κονδύλια και λέμε πώς θα δαπανίσουμε σωστά αυτά τα κονδύλια και από την άλλη πλευρά έχουμε έναν μεγάλο ευρύ κόσμο των πανεπιστημίων, ε, έναν ευρύ ακαδημαϊκό κύκλο και μας λείπει η σημαντικότερη, ο σημαντικότερος κληρίκος της αλυσίδας που είναι οι εμπειρογνώμονες. Όχι εμπειρογνώμονες για την δαπάνη των κονδύλιων, αλλά εμπειρογνώμονες και τεχνική για, ε, για το τι είναι το πιο σημαντικό στην επιστήμη, στην έρευνα, ποια ομάδα και τι είδους προγράμματα έχουν ε, μεγαλύτερες, επιτυχίες, μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό χρειαζόμαστε, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σε θέματα ε, προγράμματος της Επιτροπής, ε, όπως ε, το σημείο 37, που ε, πολύ ακροθυγώς αναφέρεται στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ κατά τη γνώμη μου έχει κεφαλαιότητη σημασία. Θέλουμε λοιπόν ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, που είναι πραγματικά κορυφαίοι στο έργο τους και φυσικά θα αμυφθούν για την εμπειρογνωμοσύνη τους και μερικοί τέτοιοι εμπειρογνώμονες θα πρέπει ε, να προέρχονται από συγκεκριμένους τομείς ε, σε, από διάφορες χώρες και ε, εδώ να έχουν επιρροή και συγκεκριμένες χώρες για την επιλογή των ονομάτων αυτών των εμπειρογνωμόνων. Επίσης, οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να υπάρχουν σε ένα σύστημα αξιολόγησης, θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα τέτοιο επιπέδων, κλιμακίων και αξιολόγησης και εκεί θα αναφέρονται συγκεκριμένα τα διάφορα θέματα ανάλογα με την αριστεία του συγκεκριμένου επιτελείου. Ανάλογα με τις δημοσιεύσεις που έχει κάνει ένα συγκεκριμένο επιτελείο, τα διπλώματα βριστεχνίας, τις διαλέξεις που έχει δώσει, τη συμμετοχή σε σεμινάρια. Αυτά θα λαμβάνονται υπόψη για το κόστος. Και φυσικά θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων. και άλλοι ομότιμοι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να αξιολογούν αυτό το έργο. Γιατί εμείς με πολύ παλιλικό τρόπο προσεγγίζουμε το θέμα της χρηματοδότησης. Λέμε πώς θα δαπανίσουμε τα κονδύλια. Αλλά κονδύλια μπορούν να δαπανίσουμε με τρόπο είτε ε, σωστό είτε λιγότερο σωστό. Θα πρέπει να δούμε πόσοι εμπειρογνώμονε πιστεύουν ότι θα πρέπει να δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια με σωστό από επιστημονική άποψη τρόπο επαναλαμβάνω, στο προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο τα ε, κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης δεν εκμεταλλεύτηκαν, δεν αξιοποίησαν όντως ε, το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο και ελπίζω στο 8ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο να έχουμε πολύ καλύτερη κατάσταση για τις χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να ανατραπεί αυτή η δυσμενή στάση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκέρεκ. Η ε, κυρία Νταλκαστίγιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι λακωνική γιατί με κάλυψαν οι προλαλήσαντες σχεδόν σε όλα τα σημεία. Νομίζω ότι εκκινώντας από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλύθηκαν πολλές προτάσεις και στην έκθεση Καρβάγιο και στην έκθεση ΟΝΤΗ για την αναθεώρηση του 7ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου, αλλά τις βλέπουμε και στη συγκεκριμένη πρόταση του κυρίου Έλλερ. Και ο κύριος Έλλερ περιλαμβάνει κάποιες από τις προτάσεις των δύο προηγούμενων εκθέσεων, Όντι και Καρβάλιο. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πραγματικά για τις άοκνες προσπάθειές του και το πολύ καλό αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε ο εισηγητής. Εγώ δεν θα επιμείνω στο αν θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ της μείωσης του άμεσου κόστους και του συνολικού κόστους ε, είτε τη συντόμευση της προθεσμίας για την επιχορήγηση σε έξι μήνες ή την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας και να ενημερώνονται τακτικά για, το, για την πορεία των αιτήσεών τους οι συμμετέχοντες. Δεν θα επιμείνω σε όλα αυτά τα επιμέρους σημεία. Θα ήθελα απλώς να κάνω δύο συμπληρωματικές παρατηρήσεις. Μία είναι προφανής γιατί είχαμε παρόμοιο πρόβλημα στο παρελθόν. Οι κανόνες συμμετοχής και η ρύθμιση της συμμετοχής γίνονται κατά την έναρξη του ορίζοντα 2020. Αυτό είναι στοιχειώδες, κάτι που δεν ίσχυσε στο παρελθόν. Έπρεπε να έχουμε ερμηνευτικές ικανότητες, ώστε όταν ε, ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος πλαισίου, δεν είχαμε ακόμη προσδιορίσει τους κανόνες συμμετοχής και χρειάστηκε να επαφεθούμε σε μια ερμηνευτική προσπάθεια. Οπότε, εδώ, είτε θα αντιμετωπίσουμε τον ορίζοντα 2020 και τους κανόνες συμμετοχής και όλα αυτά τα προγράμματα του πακέτου, είτε θα αντιμετωπίσουμε ως έναν τρόπο ε, ε, αντιμετώπιση των αναπτυξιακών πολιτικών ή οι δυνατότητες που θα μας δίνει το Ευρώπη 2020 και οι χρηματοδοτικές ε, ε, πιθανότητες θα είναι πολύ προβληματικές. Νομίζω ότι το ορίζοντας 2020 και οι συμπληρωματικές προτάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο, να εκλειφθούν ως ουσιαστικό στοιχείο του πακέτου της ανάπτυξης. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε πολύ περισσότερες δυσκολίες δημοσιονομικές. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι στρατηγική για να έχουμε καλή χρηματοδότηση για το ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο και τα συμπληρωματικά προγράμματα. Νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλλει με σημαντικό τρόπο στην ανάκαμψη της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα πρέπει να το διατρανώσουμε και με αυτούς τους όρους να γίνεται διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Να θεωρήσουμε αυτό το πρόγραμμα ως αποφασιστικό στοιχείο του πακέτου για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαδουρέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πραγματικά επιγραμματική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας τον κύριο Έλερ για το έργο του και μια και δεν μπόρεσα να το πω και χθε, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία που είχαμε. Εγώ είμαι ισκιώδη συγγήτρια για τον... Ε, μάλλον τον ευχαριστήσω γιατί είναι ισκιώδη συγγητής ε, στον κανονισμό για τον οποίο εγώ έχω την έκθεση. Τώρα, όπως είπε ο κύριος Γκλάντε, ο, ο σκιώδης ηγετής της ομάδας, αλλά και άλλοι προλαλήσαντες, είναι σημαντική η πρόταση έκθεση για τους κανόνες συμμετοχής. Στην πρόταση έκθεση με εξέπληξε ο κύριος Σέλερ γιατί είπε ότι τα άρθρα 19 και 20 θα, του κανονισμού αυτά που, αφαιρούν, αυτά που αφορούν τις συμπράξεις ε, δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, δημοσίου-δημοσίου φορέα είπε να τα ξεπεράσουμε και να πάμε κατευθείαν στους κανόνες συμμετοχής. Εγώ προτιμώ την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σημείο αυτό. Γιατί έχουμε συγκεκριμένου τομεί με βάση την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του οποίου του προσδιορίζει και όλα. Και πιστεύω ότι αυτοί οι τομεί θα πρέπει να περιγράφονται και να προσδιορίζονται και στον κανονισμό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και οι κανόνε συμμετοχή δεν θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και επίσης διαφανής. Γιατί είπαμε ότι όλες οι δράσεις του προγράμματος πλαισίου θα πρέπει να είναι διαφανείς και το ίδιο να ισχύει και στη συμπράξη είτε είναι δημοσίου, δημοσίου είτε δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. αυτό συμφωνούμε. Υπέρ της διαφάνειας και της συγκεκριμενοποίησης των κανόνων συμμετοχής. Αυτό όμως χρήζει περαιτέρω συζήτησης, γι' αυτό δεν θα μακρηγορήσω. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που σας παρουσίασε ο σκιώδης της πολιτικής μου ομάδας. Ευχαριστώ. Thank uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Έλερ για την πολύ καλή δουλειά που έκανε για τους κανόνες συμμετοχής. Όπως θα ξέρετε, έχω υποβάλει 67 συστάσεις για την απλούστευση και ήδη οι περισσότερες έχουν αναλυθεί από την Επιτροπή. Σε δύο όμω από αυτέ δεν ήταν τόσο φιλόδοξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο θα ήθελα και ο κύριο Έλλερ τι δύο αυτέ συστάσει τι έχει ενσωματώσει στην έκθεσή του. Η πρώτη αφορά το χρόνο για την δωρεά, για την επιχορήγηση ιδίως για τις μικρές δομές, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλαδή. Αυτό ευτυχώς μπόρεσε να εσωματωθεί χάρη στην ευελιξία του κ. Έλλερ. Μείωσε του χρόνου για την επιχορηγήση, για τη διάθεση της επιχορηγήσης. Και επί τα του συστήματος της καταγραφής. Η Επιτροπή προτείνει ότι οι ερευνητέ που 100% είναι αποσιωμένοι σε ερευνητικά προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ε, συμμετέχουν σε αυτό το σύστημα καταγραφή, αλλά να ισχύει για του υπόλοιπου. Αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και θα πρέπει να απλουστεύσουμε περαιτέρω τη διαδικασία. Επίσης, να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να καλωσορίσω την ε, ενσωμάτωση του ΦΠΑ ως επιλέξιμου κόστους και στο δημοσιονομικό κανονισμό έχει συμφωνηθεί αυτό και είναι ζήτημα που καίει όλους τους ευερευνητές στην Ευρώπη. Πολύ καλός λοιπόν τελικό σχέδιο της έκθεσης συμπεριλαμβάνεται. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να θυμίσω κάτι που είπε ο Άινσταϊν. Θα πρέπει όλα να γίνονται στο δυνατόν απλούστερα όσο το δυνατόν απλούστερα, αλλά όχι απλώς να απλοποιούνται. Η πραγματικότητα είναι περίπλοκη. Θέλουμε να την απλουστεύουμε, αλλά θα πρέπει να πετυχαίνουμε και την σωστή ισορροπία. Μεταξύ πραγματικότητα και απλότητα, λοιπόν, νομίζω ότι στο σωστό σημείο έχει τοποθετηθεί η έκθεση του κυρίου Έλερ. Γίνεται πιο απλή, αλλά όχι απλούστατη. Ευχαριστούμε, κυρία Καρβάλιο. Ήθελα όχι να μη σας παρουσιάσω, αλλά να σας αφήσω να τα πάρετε κατευθείαν να πείτε αυτά που θέλετε. Ο κύριος Κουάντρας. Ευχαριστώ. Χθες είπα στα γενικά μου σχόλια για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ότι ο θεμελιώδης στόχος αυτού του 8ου ερευνητικού προγράμματος πλαισίου είναι να αξιοποιηθούν καλύτερα τα κοινοτικά κονδύλια και γι' αυτό προαπαιτείται καλή διαφήμιση μεταξύ των συμμετεχόντων, μία ε, κατακήρυξη των προγραμμάτων ε, διαφανής και όσο λιγότερο γραφειοκρατική γίνεται και μία προσπάθεια ώστε η έρευνα που χρηματοδοτούμε ή συγχρηματοδοτούμε να βελτιώσει μία από τις βασικές αδυναμίες του συστήματός μας που είναι η καθυστέρηση που σημειώνουμε, η στέρηση που σημειώνουμε σε σχέση με βασικούς ανταγωνιστές μας στο πέρασμα μεταξύ της γνώσης και του προϊόντος. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη υστέρηση. Στο πακέτο που εξετάζουμε για τους κανόνες συμμετοχής και διάδοσης, σίγουρα ε, έχουμε το σημείο που επηρεάζει άμεσα την υλοποίηση των στόχων μας και το σχέδιο έκθεσης που μας υπέβαλε ο κύριος Έλλερ συνάδει με τους στόχους αυτούς προτείνοντας πολύ ε, σωστά μέτρα. Συντόμευση της ε, προθεσμία για τη χορήγηση των επιχορηγήσεων, η δημοσίευση ενός εχειριδίου, ενός οδηγού που εξηγεί τα κριτήρια της κατακύρωσης, ε, της ανάθεσης, επίσης κριτήρια με βάση με το μοντέλο και την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η έγκριση προηγούμενων προγραμμάτων. Αυτά όλα διευκολύνουν την κατάσταση. Επίσης, ε, είναι πολύ δόκιμος ορισμός των δραστηριοτήτων που είναι κοντά στην αγορά και τον αποκλεισμό κάποιων προγραμμάτων που αντιβαίνουν σε αρχές διοντολογίας ηθικής, στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του προγράμματος. Ίσως το ένα από τα πιο επίμαχα σημεία της έκθεσης του κυρίου Έλερ αφορά την κατάργηση του ενίου ποσοστού χρηματοδότησης που εφαρμόζεται για τις ε, διάφορες κατηγορίες συμμετεχόντων. Δηλαδή, αυτό το μέτρο, ο ενιαίος συντελεστής που θα απλούστευε κατά πολύ τα πράγματα, ίσως θα τα παραπλούστευε. Γι' αυτό το κατήργησε ο κύριο Έλλαρ γιατί σίγουρα μια μεγάλη επιχείρηση δεν είναι σαν μια μικρή. Ούτε ένα ερευνητικό κέντρο είναι το ίδιο με ένα πανεπιστήμιο. Και το να εφαρμόζουμε σε όλου ε, τον ίδιο συντελεστή, όντω απλουστεύει τα πράγματα, αλλά ίσω τα παραπλουστεύει. Γι' αυτό και πολύ σωστά ο κύριος Έλερ έκανε ένα σχόλιο για το θέμα αυτό και είπε να διαγραφεί αυτή η διαφοροποίηση. Πάντως ε, η έκθεση δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και αποτελεί μια εξαιρετική βάση για τη βελτίωση και την αποκατάσταση μεγαλύτερη διαφάνεια για τη διαδικασία επιλογή των διαφόρων σχέδιων και προγραμμάτων. Ευχαριστούμε κύριε Βινταλ Κουάδρα. Ο κύριο Βανίλη Σερόι Θέρμα παρακαλώ κύριε Βανίστε Ρόι, χρόνο φίδου γιατί έχουμε καθυστερήσει. Πόσα λεπτά δηλαδή. Δύο. So, I think, uh, Ο κύριος Έλερ, να ευχαριστήσω μάλλον τον κύριο Έλερ, για όλη την καλή μας συνεργασία και που άκουσε όλους τους συναδέλφους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιες παρατηρήσεις. Ανησυχώ λίγο για το γεγονός ότι εμείς προχωρούμε, ενώ μεταξύ τα κράτη-μέλη, οι χώρες δηλαδή, κάνουν περικοπές στις επενδύσεις τους. Αυτό που ίσχυε ότι ένα και ένα ίσον τρία τώρα μας οδηγεί στο μηδέν. Ένα και ένα ίσον μηδέν. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε πάλι με την εντολή που έχουμε ως Επιτροπή Ήτρε, να συζητούμε με το Συμβούλιο εμείς μπορεί να αποφασίζουμε, αλλά εκείνοι μπορεί να τα περικόπτουν όλα από την άλλη. Τι πρέπει να κάνουμε, να πιέσουμε τα κράτη, να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι σημαντικό και λείπει για την ώρα. Επίσης κάτι άλλο, η προβολή της όλης προσπαθία μας. Είναι πολλά τα ονόματα. Εγώ πρέπει να κοιτάξω πολύ χαμηλά στην ε, λίστα για να δω ποια προγράμματα είναι αυτά που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να μην ξεκινήσουμε πρώτα λοιπόν με αυτά και να έρθουν μετά τα υπόλοιπα. Μας λείπει πάρα πολύ σωστή προβολή των προγραμμάτων. Δεν τα κάνουμε σωστά τα πράγματα. Προσπαθούμε να είμαστε οι πρώτοι, να πετύχουμε κάποια πράγματα, αλλά είμαστε σχεδόν αόρατοι στην πραγματικότητα. Όχι μόνο με τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και με το κοινωνικό ταμείο και άλλα. Την έκθεση που εγώ ετοιμάζω για την εναρμόνιση και τα ποσοστά χρηματοδότηση. Νομίζω ότι λογικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση, όπως και ο κύριο Έλερ το προτείνει, αλλά τι λεπτομέρειε ίσω να τι επεξεργαστούμε. Θα ολοκληρωθεί και αυτή η προσπάθεια για να συντομεύω, σωστά τα λέτε τα περισσότερα, αλλά είναι δύο τα σημεία στα οποία πρέπει να ε, επιμείνουμε. Προβολή και να συμμετέχουν και χώρε. Διότι εάν ε, δαπανούμε λιγότερα στην Ευρώπη, δεν νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει τίποτα σε δύο χρόνια. Ευχαριστούμε κύριε Βανίστερο. Η, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Βούτσερ. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Έλερ για το σημαντικό αυτό σχέδιο έκθεση σε ό,τι αφορά του κανόνε συμμετοχή. Ευχαριστούμε που στηρίζει για κάποιε από τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίω ό,τι αφορά την απλούστευση. Οι κανόνε συμμετοχή είναι το κατεξοχήν νομικό εργαλείο που θα μα επιτρέψει να πετύχουμε αποτελέσματα στην απλούστευση και στις πολλαπλές και επανειλημμένες, ε, στα επανειλημμένα αιτήματα που έχουμε λάβει από το Ευρωκοινοβούλιο και τα κάτι μέλη ως προς την κατεύθυνση αυτή. Επειδή λοιπόν πολλά ερωτηματικά έχουν τεθεί σε σχέση με την απλούστευση, νομίζω συμφωνούν όλοι ότι χρειάζεται περισσότεροι να αρθεί το δημογραφικό άχθο για του συμμετέχοντε και να επιταχυνθούν οι χρόνια αναμονή. Επίση, να ε, μειώσουμε τι πιθανότητε ε, οικονομικών αναταραχών, διότι οι περισσότεροι ε, ουσιαστικά διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση με τα ερευνητικά προγράμματα που καθυστερούν πολλές φορές και ένα χρόνο. Και επίσης να δούμε τι γίνεται με το πρόγραμμα πλαίσιο 7 και τα σχέδια που έχουν χρηματοδοτηθεί από αυτό. Ε, θα πρέπει μετά από όλε τι συνομιλίες που έχουμε κάνει, να δούμε ότι ένα τρόπο να σταθμίζονται όλοι οι συμμετέχοντε και όλε οι δραστηριότητε από τη μια και η πρόταση τα έμεσα κόστη να αντικατασταθούν από ένα καταποκοπήν ποσό δεν επιτυγχάνει τους τρεις στόχους που θέλουμε ταυτόχρονα να επιδιώξουμε. Ένα από τα βασικά στοιχεία που αναφέρει ο κ. Σέλερ στο σχέδιο εκθέσης του είναι να παραταθεί η προσέγγιση του 7ου προγράμματο πλαισίου. Η διάκριση των ποσοστών χρηματοδότηση μεταξύ των διαφορών ιδρυμάτων, τα διάφορα μοντέλα κατά αποκοπήν ποσών με το υπάρχον πρόγραμμα είναι η προσέγγιση που σήμερα ισχύει, αλλά ήδη συζητούμε νέα ποσοστά χρηματοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν ανησυχούμε. Αν η διαφοροποίηση μεταξύ συμμετεχόντων και δραστηριοτήτων ε, συνεχιστεί, αυτό θα επιτείνει το γραφειοκρατικό άχθος. Δεν θα ε, επιταχύνουμε τους χρόνους αναμονής και δεν θα δίνονται γέρο οι επιχορηγήσει. Το ίδιο και για την πρόταση να αντικατασταθεί το έμεσο κόστο με καταποκοπήν πληρωμή. Ό,τι αφορά το χρόνο μέχρι την επιχορήγηση, είναι σημαντικό θέμα αυτό. Το ανέφερε και η κυρία Καρβάλιου. Διαπραγματευόμαστε δημοσιονομικού κανονισμού αυτή τη στιγμή και έχουμε σαφεί οδηγίε από την κυρία Γκρέσλε, δική σας συνάδελφο, ότι στον δημοσιονομικό κανονισμό δεν θα πρέπει να προβλέπονται στοιχεία για τον ε, για τους κανόνες συμμετοχής. Το ίδιο και για το ΦΠΑ και για το θέμα της, ε, των επιχορηγήσεων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τριμερής διάλογος για το δημοσιονομικό κανονισμό μεταξύ Συμβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις η περίοδος αναμονής είναι 9 μήνες για την επιχορήγηση. Δεν θα πρέπει λοιπόν μετά από τόσο μακρό σκέλη συζητήσεις να ισχύουν διαφορετικοί κανόνε για τον τομέα τη έρευνα. Αυτές είναι οι βασικές μα παρατηρήσεις για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Έλερ τα σχόλιά σας. Ε, Δύσκολο βέβαια είναι να απαντήσει κανείς τώρα σύντομα σε όλα αυτά. Θα πω δύο πράγματα και πρώτα για το γενικότερο θέμα, εάν δηλαδή υπάρχει διαφοροποίηση και αν θα οδηγηθούμε ξανά στο ε, πρόγραμμα πλαίσιο 7. Εκεί όμως το πρόβλημα δεν ήταν διαφοροποίηση, αλλά οι κανόνες. διαφοροποίηση δεν ήταν λάθος, αλλά οι κανόνες ήταν πολύ περίπλοκοι και ασαφείς. η επιχειρηματολογία της ε, Κομισιόν είναι σαν να μας λέει ότι με δύο πόδια δεν μπορούμε να περπατήσουμε, καλύτερα πάμε με ένα. Αλλά βέβαια πιο γρήγορα περπατάει κανείς με δύο πόδια. Άρα ε, καλούμαστε εδώ να συζητήσουμε λίγο περισσότερο την ουσία. Δεν θέλουμε να έχουμε δύο ανταγωνιστικά συστήματα. Σε πολλά η, Κομισιόν, η πρόταση της Κομισιόν μάλλον είναι εξαιρετικά πολιτική. Πρέπει να δούμε εάν στην εφαρμοσιμότητα, στην πράξη, πράγματι μπορεί να επιτύχει. Το Κοινοβούλιο δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ να γίνουν τα πράγματα περιπλοκότερα, έρχονται διάφορε γενικέ διευθύνσει και άλλε μονάδε τη Κομισιόν και λένε Α, να συμπεριληφθεί και εκείνο και το άλλο. Είναι πολύ ζωηρή η συζήτηση. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει συνεργασία. Αντιθέτω, αυτό που με ενδιαφέρει, αυτά μάλλον που με ενδιαφέρουν εμένα είναι ιδίω δύο πράγματα. Αφενό, η συνεπής εφαρμογή τη εκθέσεω τη κυρίας Καρβάλιο, ώστε και οι γραμμέ που ακολουθούμε να είναι καθαρές. Αυτό το έχει πράξει η Κομισιόν σε πολλά σημεία. Τα υπόλοιπα τα προσθέτουμε επειδή υπάρχει στο Κοινοβούλιο σημαντική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει υπέρ. Το δεύτερο είναι οι δημοσιονομικοί κανονισμοί. Εδώ στους financial regulations μα λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο στους κανόνες από αυτά που λένε οι financial regulations. Αυτό δεν ισχύει απόλυτα, διότι οι financial regulations οι κανόνε είναι πολύ γενική και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εξειδικεύσεις στους κανόνες. Έχουμε λοιπόν συζήτηση με τους συναδέλφους μας της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού με την έννοια ότι τα βήματα που θέλουμε να κάνουμε προς την κατεύθυνση της απλούστευσης να είναι και εξασφαλισμένα και απέναντι στο ελεγκτικό συνέδριο και απέναντι στον έλεγχο του προϋπολογισμού. Αυτά σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα διαπραγματεύσεών μας για τους financial regulations. Τώρα, δύο πράγματα ακόμη. Πρώτα, για το ερώτημα, μάλλον με ένα παράδειγμα, σχετικά με το ερώτημα ποια εξισορρόπηση πρέπει να επιδιώξουμε. Μία παρέμβαση χωρίς να κάνουμε διάκριση μεταξύ μικρόμεσων επιχειρήσεων και βιομηχανίας. Με την έννοια ότι χρειάζονται 4-6 εβδομάδες για να κριθεί μία αίτηση, να διαπιστωθεί δηλαδή εάν πρόκειται για αίτηση μικρής μεσαίας επιχειρήσης ή όχι. Από άψη οικονομική είναι απολύτως παράλογο να έχουμε ένα ενίο συντελεστή παρέμβασης. Χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση μικρή και μεσαία επιχείρηση από τη μεγάλη βιομηχανία. Αυτό είναι σαφές. Αυτό όμως που λέει η Κομισιόν ότι χρειάζεται 4 6 εβδομάδες για να αποφασίσει αν πρόκειται για μικρή μεσαία επιχείρηση ή για βιομηχανία. Το ερώτημα είναι να μην κάνουμε πλέον τη διάκριση μεταξύ ΜΜΕ και βιομηχανία, Διότι αλλιώ παρέρχεται αυτό το περιθώριο των 6 εβδομάδων, ούτως ή άλλως. Να πούμε ότι από άψη οικονομική βεβαίω πρέπει να γίνεται η διάκριση μεταξύ ΜΜΕ, μικρή και μεσαίες επιχείρηση βεβαιω δηλαδή, και βιομηχανίας, αλλά η διακριση μεταξυ μμε μικρη και μεσαια επιχειρηση δηλαδη και βιομηχανια αλλα η κομισιον να μην χρειάζεται 6 εβδομάδε, αλλά να το καταφέρνει σε λιγότερο περιθώριο. Δεν νομίζω ότι κάθε διαφοροποίηση είναι ο εχθρός της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Χρειάζεται να γίνεται η απαραίτητη διαφοροποίηση έτσι ώστε να δώσουμε οικονομικά τα ορθά κίνητρα και ταυτόχρονα να φροντίσουμε ώστε τα πράγματα να παραμένουν απλά. Αυτή λοιπόν η εξισορρόπηση θα είναι και το καθήκον μας τους επόμενους μήνες. Είναι ενδιαφέρον που ακούμε για πρώτη φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια εμπειρικά στοιχεία. Προηγουμένως δεν είχαμε μπροστά μας παρά ένα black box, ένα μαύρο κουτί. Δεν ξέραμε καθόλου τι ε, δεδομένα υπήρχαν μέσα. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο είναι επαρκώς ευφυές και έχει και διάθεση συνεργασίας με την Κομισιόν. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε εμπειρικές ενδείξεις, όχι απλά πολιτικές δηλώσεις. Και η Κομισιόν λοιπόν θα πρέπει να προσέξει δεν σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θέλει να επανέλθει στο πρόγραμμα πλαίσιο 7, ενώ η Κομισιόν θέλει κάτι το πολύ φιλόδοξο. Έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα η Κομισιόν το οποίο είναι σωστό ό,τι αφορά του προσανατολισμού του, αλλά μα έρχεται μια ανακοίνωση μετά την άλλη. Και στι ανακοινώσει αυτέ σχολιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι ίδιε τι νομοθετικέ προτάσει. Μιλεί για διεθνοποίηση και ούτω καθεξή. Εγώ λοιπόν δεν ανησυχώ δεν θεωρώ ότι ισχύει η μομφή ότι θέλουμε να επανέλθουμε στο FP7, στο ε, πρόγραμμα πλαίσιο 7. Αλλά περισσότερο μας απασχολεί το ερώτημα εν ώψη των σημαντικών δημοσιονομικών προβλημάτων πώς θα πετύχουμε πρώτο μια μόχλευση, δηλαδή με τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας να μπορέσουμε να ενισχύσουμε όσο γίνεται περισσότερο την έρευνα και την ανάπτυξη, χωρίς να πούμε στις στατιστικές δυσκολίες ότι θα, θα λένε ότι δίνουμε περισσότερα χρήματα στη βιομηχανία που θα έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή της βιομηχανίας τότε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη μόχλευση. Θέλουμε λοιπόν απλούστευση, μόχλευση, να ρυθμιστούν τα πράγματα έτσι που να μπορεί να τα διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι δεν είμαστε και αντίπαλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αναμένω με ήρεμο πνεύμα την συζήτηση που δεν θα είναι καθόλου ιδεολογική. Και αυτό ήταν άλλωστε το ικανοποιητικό στο πιο πρόσφατο παρελθόν, ότι δηλαδή μπορέσαμε μαζί να καταλήξουμε σε συμβασμού. Και αυτό αναμένω να γίνει ακόμη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εσά κύριε Έλερ. Σε λίγο βέβαια θα αναγκαστούν να φύγουν οι διερμηνεί και θα κάνουμε διάλειμμα. Έχουμε όμως ακόμη 10 λεπτά. Με διερμηνία 10 λεπτά για την τελευταία έκθεση του σημερινού πρωινού. Πριν όμως από αυτό, να σας πω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 27 έκτους στις 12 το μεσημέρι. Προχωρούμε τώρα με ταχύτητα στην επόμενη έκθεση, Κάλφιν. Ο ίδιος ο κύριος Κάλφιν ε, συμμετέχει σε συνάντηση με τον πρόεδρο σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμως όσα είχε να πει τα είπε χθες. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε αμέσως τους σκιώδεις εισηγητάς και ο πρώτος είναι του Λαϊκού Κόμματος. Ο κύριος Αδαλμπάρα. Ευχαριστώ. Δύο λόγια μόνο να κάνω κάποια σχόλια στα πλαίσια αυτής της ανταλλαγής απόψεων. Καταρχήν, όταν μιλούμε για την αναθεώρηση της ε, συγκεκριμένης οδηγίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μιλούμε για την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών, όχι για την πρόσβαση στα έγγραφα. Προσοχή λοιπόν, μιλούμε για τη χρήση των πληροφοριών του δημόσιου τομέα και όχι για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα. Θα ήθελα να τονίσω κάποιες από τις προκλήσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε και την ανάγκη τροποποίησης, αναθεώρησης της ως οδηγίας. Καταρχήν, οι δημόσιοι φορείς δεν είχαν γνώση την πιθανότητα αυτής της επαναχρησιμοποίησης. Δεν υπήρχε σωστή ενημέρωση και θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία της διοίκησης ως προς το θέμα αυτό. Επίσης, χρειάζεται κάποια εναρμόνιση των κανόνων που ισχύουν στα κράτη-μέλη, που είναι διαφορετική και επίσης εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο η ισχύουσα νομοθεσία, η σχετική οδηγία. Θα πρέπει να αποκατασταθεί μια ομοιομορφία λοιπόν. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της οδηγίας τώρα, της αναθεώρησης της οδηγίας. Καταρχήν, το πεδίο εφαρμογής αυτής της νέας χρήσης. Με την αναθεώρηση περιλαμβάνονται τα μουσεία, τα βιβλιο... οι βιβλιοθήκες και τα πανεπιστήμια στις πληροφορίες στο δημόσιο τομέα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Δεύτερο σημαντικό σημείο, η χρέωση. Τι θα τι ε, τέλη θα καταβάλλονται ή αν θα είναι δωρεάν αυτή η επαναχρησιμοποίηση. Βασικό στοιχείο λοιπόν η χρέωση. Θα πρέπει να δούμε ποιο, ποιο είναι το περιθωριακό κόστος γιατί δωρεάν επαναχρησιμοποίηση δεν σημαίνει ε, νέα χρήση τελείως ε, χωρίς κόστος. Επίσης, ε, μερικές φορές δεν είναι μόνο δημόσιοι φορείς. Είναι και ιδιωτικοί φορείς που καλύπτονται από ένα δημόσιο προϋπολογισμό. Οπότε και τα προϊόντα που παράγουν, οι πληροφορίες θα πρέπει να εμπίπτουν. Να μην περιορίσουμε λοιπόν αυτούς τους προϋπολογισμούς ή να μην αυξήσουμε το έλλειμμα της δημόσιας διοίκησης. ώστε να παίρνει και το δημόσιο ένα τμήμα αυτών των τελών που θα καταβάλλονται από την πόλη του προϊόντος. Τώρα, πώς θα χρησιμοποιούνται αυτά τα μεταδάτα, ποιο είναι το λογικό format για την επαναχρησιμοποίηση των πληροφοριών. Το θέμα του format είναι πολύ σημαντικό. Ο μορφότυπος. Επίσης, ποια θα είναι η εποπτική αρχή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη σύσταση ενός ανεξάρτητου φορέα. Κατά τη γνώμη μου, αν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των θεσμικών οργάνων των κρατών μελών, των αρμόδιων αρχών, δεν χρειάζεται ένα καινούριο σώμα, μια νέα ανεξάρτητη αρχή. Πάντως αυτό που χρειαζόμαστε είναι πραγματικά αμερόληπτη και ανεξάρτητους φορείς, ώστε να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότητα, θεμητός ανταγωνισμός και διαφάνεια μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα, ώστε να έχουμε καλή νέα χρήση αυτών των πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Και τονίζουμε ότι υπάρχει εδώ μεγάλο δυναμικό που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να αυξηθούν τα ωφέλη και για το δημόσιο και για τον ιδιωτικό φορέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βάλιαν μου ζήτησε να σας διαβάσω το εξή κείμενο. Πιστεύω όλοι συμφωνώ που πρέπει να θεωρηθεί αυτή τη στιγμή η οδηγία και είναι σωστή η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το νέο νομοθέτημα θα πρέπει να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και οικονομικά ωφέλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας. Όμως πρέπει να διαβεβαιωθούμε ότι αυτή η οδηγία όχι μόνο θα πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά ε, θα πρέπει να βελτιωθεί ως προς την πρόταση της Κομισιόν που είναι υπερφιλόδοξη. Θα πρέπει το πεδίο να συμπεριλάβει και άλλους δημοσίους φορείς, αλλά να δώσουμε μεγάλη προσοχή και στο πώς θα υλοποιούνται οι νέες διατάξεις. Ιδάλλως, υπάρχει κίνδυνος κάποια ιδρύματα τελικά να μην διαθέτουν καμία πληροφορία, έστω πολύ λίγε, κάτι που θα κυρώσει και το σκοπό αυτή τη αναθεώρηση. Επιπλέον, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στι ενδεχόμενε αρνητικέ συνέπειε τη δημοσιοποίηση δεδομένων. Εδώ σκεφτόμαστε την περίπτωση κατάχρηση προσωπικών δεδομένων που θα μπορούσε να προκύψει με την ε, διευκόλυνση τη πρόσβαση της πληροφορίας. Θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα εχέγγυα ώστε οι ενδεχόμενη αύξηση της, των απειλών κατά τη ιδιωτικού βίου να αποφευθούν εφόσον αρχίσει να υλοποιείται η οδηγία. Θα πρέπει να εξεύρουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ φιλόδοξου πεδίου εφαρμογής και ενός ρεαλιστικού νομοθετήματος που θα βελτιώσει τη διαφάνεια χωρίς να την εμποδίζει και τον δίκαιο ανταγωνισμό αλλά και την ιδιωτικότητα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Η έκθεση είναι πρόσδεκτη και χαίρομαι που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να συζητήσουμε τη δημοσιοποίηση δεδομένων εδώ. Είναι πολύ καλή βάση η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χαίρομαι ιδιαίτερα που κάποιοι εδώ συμφωνούμε με αυτήν την θέση. Είναι καλή βάση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διευκόλυνση πρόσβαση σε περισσότερο υλικό και στη συμπερίληψη περισσότερων τομέων. Θα πρέπει βεβαίω να οριστούν και το τι είδου ενέργειε θα μπορεί κανεί να επιτελέσει με αυτό το υλικό. Εάν σκεφτούμε τι ενώσει πολιτιστικών, το τι υλικό έχουν στα χέρια του, τι βιβλιοθήκε στα πανεπιστήμια, καλύπτονται και αυτά. Όμω, ξεχνάμε ταυτόχρονα ένα σημαντικό στοιχείο του δημόσιου τομέα, δηλαδή τι δημόσίε υπηρεσίε αυτές καθ' αυτές εδώ και έναν αιώνα οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν πληρώσει και για ραδιοφωνικούς σταθμούς και πολλά που έχουν καταφέρει οι πολιτιστικές αυτές ενώσεις. Οι τηλεοπτικές σειρές λόγου χάρη ήταν κάτι που βοήθησε πολύ την προσωπική ανάπτυξη της γενιάς των γονών μου λόγου χάρη. Τα πράγματα εντωμεταξύ έχουν αλλάξει. Καθυστέρησε λοιπόν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάπως, ιδίως ό,τι αφορά τους πιο ηλικιωμένους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε ένα σύστημα, χωρίς να περάσει μια δεκαετία διαπραγματεύσεων για να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το τι θα γίνει με τα τρίτα μέρη στην περίπτωση αυτή και βεβαίως να αποφύγουμε τα προβλήματα όταν μιλάμε για τις εταιρείε ιδιωτικών υπηρεσιών. διότι εκείνοι και ξέρουν πού βρίσκονται τα πνευματικά δικαιώματα και κάποια από αυτά τα κατέχουν. Είναι σημαντικό λοιπόν κοινωνικό ζήτημα. Έχω πολλούς φίλους που βλέπουν τηλεοπτικές σειρές στο τέλος της δεκαετίας του 80. Αυτό αφορά φίλους και γνωστούς γονείς, όχι μόνον εμένα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε με περισσότερες φιλοδοξίες και εμείς από την πλευρά μας για την πρόταση της Επιτροπής. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι οι τηλεοπτικές σειρές του 80 είναι μια θετική πολιτιστική συνεισφορά. Σας ευχαριστούμε όλους. Επόμενη συζήτηση για το θέμα αυτό. Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ τους διερμηνείς.